Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Αγαπητοί μέλη, αγαπητοί ομιλητέ, κυρίε και κύριοι, με μεγάλη χαρά σα καλωσορίζω στην δημόσια αυτή ακρόαση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στα χρηματοδοτικά δικαιώματα στην Ουγγαρία. Η... Γίνεται εγγραφή των ομιλιών αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης 14ης Νοεμβρίου να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία στις αρχές του 2017. Στη συνάντηση της 16ης Ιανουαρίου το Προεδρείο έδωσε την έγκρισή του να λάβει χώρα αυτή η συνάντηση και στις 24 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος Ταγιάννη ενημέρωσε για την απόφαση αυτή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι συντονιστές της ΛΥΜΠΕ συμφώνησαν την ημερησία διάταξη καθώς και τα ονόματα των ομιλητών με γραπτή διαδικασία. Η σημερινή ακρόαση αποφασίστηκε από τους συντονιστές και ε, ε, θα φροντίσω έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των πολιτικών ομάδων και τον τρόπο διεξαγωγής. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ομιλητές για 10 λεπτά θερμή παράκληση σε αυτό που θέλω να σας πω. Τα δέκα λεπτά είναι ε, ο ακριβής χρόνος αγόρευσης. Δεν είναι ο συνιστόμενος χρόνος αγόρευσης. Θα δείτε στη μικρή οθόνη μπροστά σας πόσα λεπτά σας απομένουν ακόμα. Μόλις τελειώσει το διάστημα αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσετε άμεσα κι εσείς. Αυτό βεβαίως είναι θέμα δικαιοσύνης, αλλά οφείλεται και στο ότι ακολουθούν ψηφοφορίες αμέσως μετά από αυτή την ακρόαση. Συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε παραχωρήσεις σε κανένα θερμή παράκληση. Μη ζητήσετε κάτι περισσότερο, δεν θα γίνει δεκτό. Εγώ προσπαθώ να είμαι ευγενή, απλά και μόνο προσπαθώ να εξηγήσω το πώ θα διεξαχθούν σήμερα τα πράγματα. Βεβαίω είστε πρόσδεκτοι αν θέλετε να μιλήσετε λιγότερο από 10 λεπτά. Μιλάμε για το μάξιμο που πρέπει να είναι 10 λεπτά. Μετά από αυτό θα ήθελα να έχω τη βεβαιότητα ότι υπάρχει επαρκή χρόνο για ερωτήσει. Οι μπορούν να θα πρέπει να διατυπωθούν σε 1,5 το πολύ 2 λεπτά για να μπορέσουν να τύχουν και κάποιες απάντηση. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστείτε απόλυτα το χρόνο αγόρασης. Ο, ο των ομιλητών είναι εκτενής, παρακαλούμε να σεβαστείτε τα χρονικά όρια. Θα πρέπει να τελειώσουμε εντός των δύο ωρών που μας έχουν δοθεί. Δεν μπορούμε όμως να ε, μιλήσουμε πέραν αυτού του, συνδυάσουμε πέραν αυτού του διαστήματος γιατί έχουμε ψηφοφορίες. Επιτρέψτε μου να περάσω στον κατάλογο των ομιλητών και να ξεκινήσω με τον κύριο Ταγιάννη. Δεν θα κάνω εκτενείς εισαγωγές. Ο δόκτωρ Τροτζάνη λοιπόν, ο δόκτωρ Τροτζάνη. Κύριε Τροτζάνη, καλώς ορίσατε. Ε, παρακαλώ, πάρτε το λόγο για να μας μιλήσετε για 10 λεπτά όπως είπαμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Καταρχάς επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας προκειμένου να μιλήσουμε για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε στην αίθουσα Αγίου Ζανφωτών, ο οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση τη κομμουνιστική δικτατορία. Θα ήταν σκόπιμο να θυμίσουμε ότι στι 25 Φεβρουαρίου Θυμηθήκαμε τα θύματα του κομμουνισμού. Σήμερα βρισκόμαστε στη ζηλευτή κατάσταση να ζούμε σε μια δημοκρατία όπου η αντιπαράθεση των ειδών, η συζήτηση είναι ελεύθερη και επιθυμητή και εκταία. Το Συμβούλιο Υπουργών μου ζήτησε να εκπροσωπήσω την Ουγγαρία μέσα σε αυτή την Επιτροπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα εκπροσωπώντας ε, ε, την Ουγγαρία και θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή. Ως πρέσβης στο Παρίσι μπόρεσα να παρακολουθήσω του σύνεγγυς ε, τη συζήτηση σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα της Ουγγαρίας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ήδη από εκείνη την εποχή ε, η ε, κατόπιν πρόταση της ουγγρικής κυβέρνησης υιοθετήθηκε κατά ε, κατάλογος των ανθρωπίων δικαιωμάτων. Αυτό δείχνει σαφώς ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας είναι πάντοτε ανοιχτή στο διάλογο προκειμένου να διευκρινίσει τη θέση της. Χάρη σε αυτή την επικοδομητική προσέγγιση μπορούσαμε να εξετάσουμε όλα τα έγγραφα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε μια φάση μεγάλης αβεβαιότητας. Υπάρχει η κρίση του ελληνικού χρέους, η τρομοκρατία, το Brexit. Είμαστε ενώπιον αλλαγών. Τα κλασικά ευρωπαϊκά κόμματα θα πρέπει να δώσουν σαφείς και αποτελεσματικές απαντήσεις παραπάνω προκλήσεις. Θα ήταν σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ότι φέρουμε μεγάλη ευθύνη. Η συμβολή της κοινίας των πολιτών είναι ιδιαίτερα ευπρόσθεκτη από τη στιγμή που ο διάλογος μεταξύ των κυβερνήσεων, των θεσμών και των ΜΚΟ είναι αναγκαίο. Θα πρέπει να υπάρξει μια διάκριση μεταξύ του ρόλου που διαδραματίζουν οι διάφοροι φορεί από τη στιγμή που ε, δεν θα πρέπει να αρνηθούμε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ε, ε, τι πάει να πει νομιμότητα ήθελα να υπογραμμίσω στις συγκεκριμένου προβληματισμούς. Η κρίση, η μεταναστευτική κρίση προβληματίζει ιδιαίτερα την Ουγγαρία και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατάσταση της Ουγγαρίας, η κατάσταση είναι σοβαρή. Αυτά είναι θέματα που εξετάστηκα από την ε, Ουγγαρία και προβλημάτισαν πάρα πολλές χώρες μέλη σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των κρατών μελών και είναι πράγματα που μας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Είναι σαφές ότι η κατάσταση αυτή πλήττει τις ελευθερίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουγγαρία λαμβάνει σοβαρά την υποχρέωσή της να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα το 2015 ακούστηκαν πολλές κριτικές απέναντι στην Ουγγαρία, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι η κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζεται στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε περήφανοι που μπορέσαμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την αλλαγή νοοτροπίας. Τώρα θα ήθελα να αναφέρω μια μικρή φράση του κύριου Τόμας Δεμαγέρ, Υπουργού Εσωτερικών, που έγραψε στον κύριο Τίμερμαν και είπε ότι για να καταπολεμήσουμε την ε, λάθρομετανάστευση και το, τη διακίνηση μεταναστών, η Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει ε, σχέσεις με τις τρίτες χώρες προέλευσης ή διαμετα, ε, διέλευσης, ε, καθώς και με την υπηρεσία για τους πρόσφυγες ε, και διάφορες διεθνείς οργανώσεις. Ε, το Υπουργείο Εσωτερικών ε, δίνει μεγάλη σημασία σήμερα στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και στο λαθρεμπόριο μεταναστών. Μία από τις προκλήσεις επίσης είναι να διευκρινίσουμε κάποιες έννοιες, ε, οι οποίες ακούγονται όταν μιλάμε για τη μεταναστευτική κρίση. Βλέπουμε ότι ορισμένοι μπερδεύουν τους οικονομικούς μετανάστες με τους πρόσφυγες ε, ή ένα Σύριο από το Άλπο ε, με έναν Μαροκάνο μετανάστη. Επίσης, Σύγχυση προκαλεί η έννοια τη ασφαλούς τρίτη χώρα. Πρέπει να ξέρουμε ότι κάποια ε, κράτη-μέλη δεν θεωρούνται σίγουρε χώρε. Ε, ενώ παραδείγματο χάρη η Τουρκία ε, είναι μια σίγουρη χώρα. Οι Ευρωπαίοι ε, διερωτώνται γιατί πολλοί από αυτού που φτάνουν στο χώρο Σέγγεν μετά ε, τη διέλευση διαφόρων σίγουρων χωρών ε, δεν υποβάλλουν την αίτηση για το καθεστώς του πρόσφυγα παρά μόνο σε λίγες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στη Γερμανία. Θεμητό ερώτημα. Η Ουγγρική κυβέρνηση ε, σε αυτή την νομοθετική της ε, προσπάθεια που κάνει ε, καθοδηγείται από, την, από το μέλημα να προστατεύει το πληθυσμό τη, ε, του πληθυσμού των κρατών μελών της τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει ταχύτατη και αποτελεσματική επεξεργασία τη αίτηση και να γίνει σεβαστό το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όμω, ε, όλα τα κάτι μέλη δεν έχουν του ίδιου στόχου. Παραδείγματο χάρη, συμμετείχα στο, Υπουργείο, στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη, όπου δεν έγινε καμία συνεδρίαση χωρί να συζητήσουμε τα θέματα τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση. Το ίδιο ε, συνέβη και στο, ε, στη συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών, όπου τα θέματα προστασία του χώρου Σέγγεν είναι ένα μόνιμο ε, θέμα. Επιτρέψτε μου τώρα να σας επιστήσω την προσοχή σε μια μορφή παραβίασης ενός θεμελιώδους δικαιώματος που δημιουργεί πολλές ανησυχίες στα κράτη-μέλη που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004. Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσφατα υιοθέτησαν νόμους που εμποδίζουν την ε, ελευθερία του επιχειρήν που εγγυάται το άρθρο 16 της Χάρτας ή και η Συνθήκη. Η απόσπαση των εργαζομένων δημιουργεί ε, ε, εμποδίζεται λόγω πολλών διακριτικών ε, στάσεων και νομοθεσιών. Πολλοί, πολλοί οικονομικοί φορείς μου δημιούργησαν, μου εξήγησαν τις προσωπικές τους δυσκολίες. Ε, και όμως υπάρχει η χειρότατη σιωπή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων απέναντι σε αυτή, την παραβίαση. Ε, επίσης πρέπει να δούμε και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Ε, στις, εδώ, στη συζήτησή μας, έχουμε προσκαλέσει διάφορες οργανώσεις. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει να αντιπαρατεθούν ιδέες και όχι δόγματα εδώ. Δίνουμε μεγάλη σημασία σε ένα τέτοιο διάλογο στα πλαίσια της ομάδας εργασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου στο εσωτερικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου που κάποιες από τις οργανώσεις που είναι παρούσες εδώ ε, απέχουν μονίμως από αυτή τη δουλειά ε, κι όμω η, Ευρωπα... η Ουγγρική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το διάλογο. Ε, και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει στο... στη Βουδαπέστη, ορίστε, ερχόμαστε στη Βρυξέλλη για να το εξασφαλίσουμε. Να σα ε, παρουσιάσω του συναδέλφου που είναι ειδικοί για τα θέματα τη μετανάστευση. Ε, Ζούζαν Βεκ, ε, Γενική Διευθύντρια του Γραφείου Μετανάστευση τη Ουγγαρία, Κριστιαν Κετσμάρ, ε, Υπουργό ε, Υπεύθυνο για τι Ευρωπαϊκέ Υποθέσει, ε, που ανήκει στο Υπουργείο ε, Δικαιοσύνη. 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Έκανα. Ο κύριο Κέτσμαρκ, που είναι αρμόδιος υπουργό για τι Ευρωπαϊκέ υποθέσει και η κυρία Σουζάννα Βέγ, που είναι ε, γενική διευθύντρια του Γραφείου Μετανάστευσης Ουγγαρία. Ο κύριο Μίκλο σαν το επικεφαλής του Κέντρου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, έχει το λόγο για 10 λεπτά. Ε, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Θα προσπαθήσω και εγώ να τηρήσω το χρονικό όριο. Επιτρέψτε μου, συνεπώς, να αναφερθώ σύντομα στην Ουγγαρία, τη λεγόμενη κατάσταση στην Ουγγαρία αν και είναι μια κατάσταση που δεν σχετίζεται μόνο με την Ουγγαρία, αλλά με τη δημοκρατία γενικότερα. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να καταστήσω πολύ σαφές πως παρόλα στις άλλες εγχώριες και διεθνείς ανησυχίες, η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα συνεχίζουν να υπάρχουν πλήρως σε λειτουργικό επίπεδο στην Ουγγαρία. Το Σύνταγμα, το κύριο συστατικό της, αστυνομία, της δημοκρατίας, το 2011 ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο με, σε μια διαφανή δημοκρατική διαδικασία Φυσικά και υπάρχουν διάφοροι τρόποι λειτουργία τη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε υπό συνθήκε έλλειψη του κράτου δικαίου πω μπορούμε να έχουμε έναν ξεκάθαρο ορισμό. Υπήρξαν αλλαγές από το συνταγματικό δικαστήριο, αλλά σε άλλες χώρες έχουμε διαφορετική κατάσταση από ότι σε εμάς, παραδείγματος χάρη στη Σουηδία, στην Ιρλανδία, στην Ουγγαρία, η κατάσταση είναι διαφορετική από ό,τι στη Γαλλία που είναι σαφής που είναι σαφώς δημοκρατία, όπου η εισαγγελία... Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία που υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη και τα οποία είναι κοινέ ευρωπαϊκές αξίες. Είναι οι ελεύθερες εκλογές και ο χωρισμός των εξουσιών ε, που θα πρέπει να εγγυώνται στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, όπως ε, εγγυάται και η Ουγγαρία, το γκρικό κράτος, ε, σε τοπικό και σε ε, γενικό, ε, κρατικό επίπεδο γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια εκλογές. Ε, έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση, το εκλεστικό όργανο, ε, λειτουργεί εντελώς χωριστά από το Κοινοβούλιο. Ένας βασικός νόμος στην Ουγγαρία, αντίθετα από το προηγούμενο Σύνταγμα της Ουγγαρίας, στην παράγραφο 1 του, του άρθρου C, λέει ότι η λειτουργία του, του κράτους θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών. Ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελεύθερων εκλογών και διαχωρισμού των εξουσιών, η υλοποίηση των και προώθηση των διαφόρων τεχνικών ε, μηχανισμών και λύσεων που αφορούν διάφορους φορείς και όργανα ε, του, κρατικού μηχανισμού ακολουθεί τις νομικές παραδόσεις της χώρας μας. Ε, στο 4-3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγεται ότι η Ένωση θα πρέπει να σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών που ε, εγγράφεται ε, στις δομές τους, στην πολιτική τους, στο σύνταγμά τους, στην κυβέρνηση και, στην τοπική, και στις λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εφόσον συζητάμε για τη δημοκρατία, στην πραγματικότητα έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις για την κυριαρχία, αλλά όχι για τη δημοκρατία. Δεν είναι δεν συζητάμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Απλώς ε, υπάρχουν ε, συγκρούσεις ιδεολογικές ε, για το τι είναι εθνική κυριαρχία στα κράτη-μέλη ή για το πώς θα πρέπει να διαιρεθούν οι αρμοδιότητες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Ε, πρέπει να δώσουμε επίσης έμφαση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κράτος. Δεν υπάρχει ε, ευρωπαϊκός δήμος και επομένως δεν έχει κυριαρχία. Μόνο τα κράτη-μέλη έχουν εθνική κυριαρχία. Ε, όπως λέει και το Ουγγρικό Σύνταγμα, η Ουγγαρία ασκεί μόνο κάποιες από τις αρμοδιότητές τους που απορούν, αρέουν από αυτή τη λογική της κυριαρχίας. Ε, και μέσω των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ε, υλοποιούνται άλλες ελευθερίες. Βεβαίως υπάρχουν και άλλε έννοιε που συνδέονται με την έννοια της κυριαρχίας και το πώς θα πρέπει να ερμηνευτεί ή να αναδιαρθρωθεί. Από τη μία, η έννοια τη υπερεθνική τη υπερεθνικής ευρωπαικη ένωσης, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες ή θα πρέπει να έχει και αποκλειστική ε, κυριαρχία ει βάρος των κρατών μελών. Ε, να έχει και το δικαίωμα να ερμηνεύει και να ε, εφαρμόζει ε, κράτος δικαίου ή θεμελιώδη δικαιώματα και να τα επιβάλλει στα κράτη-μέλη. Ε, αυτό είναι ε, φονταμεταλισμός ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, πολιτική ορθότητα κτλ. Και βεβαίω έτσι μειώνται οι εξουσίε των κρατών μελών. Ε, Υπάρχουν άλλε έννοιε όπου λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εργαλείο. Άλλη, άλλη ιδεολογία αυτή. Ε, και μόνο τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να έχουν αρμοδιότητε ε, που απορρέουν από τη δική του εθνική αρχή για να διαμορφώσουν το νομικό περιβάλλον που συνδέεται με την συνταγματική του ταυτότητα, όπω παραδείγματο χάρη ε, το ρόλο του συνταγματικού δικαστηρίου, του γενικού εισαγγελέα ή οι διαδικασίε οι οποίες ε, συνδέονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Φυσικά ξέρω ότι είναι προφανές ότι αυτή είναι μόνο η αρχή μιας ε, ευρύτερης αλλαγής γύρω από τη φύση και την μορφή της δημοκρατίας, ε, την έννοια των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και όλα αυτά συνδέονται με την ε, κυριαρχία. Είναι σαφές επίσης ότι η πολιτική και νομική μάχη ανάμεσα αυτούς που θέλουν υπερεθνικές λύσεις για όλη την ανθρωπότητα και εκείνους οι οποίοι θέλουν την εθνική ταυτότητα ε, που συμπεριλαμβάνει και, εδώ, και, τον, και την ερμηνεία των θεμελιώδων δικαιωμάτων ε, είναι κάτι οποίο δεν αφορά μόνο την Ουγγαρία αλλά όλη την Ευρώπη και όλο το δυτικό ημισφαίριο όπως ξέρουμε. Επομένως, ε, νομίζω ότι οι πιο ενδιαφέρουσες μέρες της ζωής μας μας περιμένουν. Έρχονται όπου να είναι. Ευχαριστώ και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Τότζο Γκάρντος, ερευνητή από το Amnesty International. Thank you very much. Good afternoon, ladies. and Ευχαριστώ. Καλό σα απόγευμα, κυρίε και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσά σα σήμερα. Θα ήθελα να σα πω ότι η Amnesty International ε, προβληματίζεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία στο παρελθόν. Ε, Μα προβλημάτιζαν οι πρακτικές σε διάφορες περιοχές που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά την απολαβή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμπιστία μίλησε για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για τι τροπολογίε που αφορούν βασικά δικαιώματα. Είμαστε κατά της εισαγωγής νόμων χωρίς να υπάρξει προτέρα διαβούλευση και γενική συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν τρία θέματα που θα ήθελα να δείξω. Το, το πρώτο αφορά ένα μήνυμα προς όλους. Έχουμε κρούσει τον κόδωνα κινδύνου και ζητήσαμε να γίνει ένας ορισμός ε, των ε, μειονοτήτων. Τα μέτρα αυτά επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Γινόμαστε μάρτυρες ε, αλλαγών στο Σύνταγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, ε, εκστρατείες που αφορούν επιπλέον περιορισμούς του δικαιώματος στην άμβλωση. Η κυβέρνηση πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες για να προχωρήσει τα δικά του προγράμματα και καθιστώντας τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη για αυτούς τους ανθρώπους. Ο ίδιος ο Υπουργός άρχισε να ενοχλεί τις, ε, τις οργανώσεις ε, ε, ΜΚΟ. Τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση έδειξε ιδιαίτερα η σε ό,τι αφορά τους ε, Θήγκανους, ε, τους, τους, τους ε, Ρωμά, τους Μουσουλμάνους κτλ. Το κοινοβούλιο αυτό και η επιτροπή αυτή ξεκίνησε μία έρευνα και προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς κάνει η Ουγγαρία. Οργάνωσε ακροάσεις, η Διεθνής Αμνηστία ενδιαφέρεται για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνεχίζει να θέτει ερωτήσεις, απαιτώντας το σεβασμό των υποχρεώσεων όλων. Πάρα πολύ συχνά θα πρέπει να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που βρίσκονται περιθωριοποιημένοι. Το επίπεδο προστασίας ε, έχει ε, μειωθεί κατά πολύ. Οι νομικές ε, βεβαιότητες αφισβητούνται από την κυβέρνηση. Την προηγούμενη εβδομάδα η ε, κυβέρνηση και λέει International εξέδωσε ψευδείς εκθέσεις. Εμείς περιμένουμε ότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερος εκπορισμός. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μήνυμα που θέλω να σας στείλω είναι αφορά τον κατεπήγοντα χαρακτήρα του θέματος. Την ώρα που εμείς βρισκόμαστε εδώ, οι, πάρα πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες εξωθούνται στα σύνορα. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κάθε κατανόηση, κάθε ήκτο για αυτούς που εγκαταλείπουν τις αιστείες τους. Από την άλλη πλευρά δεν ε, τους ε, επιτρέπει να κάνουν κάτι. Δεν ε, αναλογίζεται τις εθνικές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει κάθε ευκαιρία να κάνει κάτι για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών. Η κυβέρνηση δεν δέχεται τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών. Από την άλλη πλευρά, πολλά ε, παιδιά, πάρα πολλοί πρόσφυγες βρίσκονται καθυλωμένοι σε ένα σημείο λόγω των προωθήσεων. Η γενική αυτή προσέγγιση οδηγεί σε μια σειρά από προβλήματα στα σύνορα. Δεν θα πρέπει να κάνουμε λάθος. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να θεωρηθεί η Ουγγαρία η χειρότερη δυνατή επιλογή για τους ετούντες άσυλο. Η Ουγγαρία δεν σέβεται τις υποχρεώσεις, τους, τις υποχρεώσεις της. Παράλληλα, η κυβέρνηση λέει ότι οι μετανάστες αποτελούν απειλή στην ασφάλεια της Ουγγαρίας. Πάρα πολλοί συνδέουν τους πρόσφυγες με την τρομοκρατία στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις έχουν δαπανίσει υπέρογκα ποσά. Τα ποσά αυτά δεν είχαν σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη προστασία για όλους. Αντίθετα, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν αντικείμενο ακόμα πιο ακραίων συμπεριφορών. ο ορισμός που δίνεται της τρομοκρατίας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η διεθνή Αμνηστία είναι ιδιαίτερα προβληματισμένη με αυτό το θέμα. Αυτό ακριβώ συνέβη στον Αχμετζέτσε, ένα Σύριο ο οποίο καταδικάστηκε άδικα το 2016 για εγκληματικές ενέργειες και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση αποτελούσε μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας προσφύγων και μεταναστών. Σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται, ε, αυτό που έκανε ο Αχμέτ είναι ότι ζήτησε ένα μεγάφορο, μεγάφορο και ζήτησε, έριξε τρία αντικείμενα ε, προς τους ε, αστυνομικούς. Στην πραγματικότητα ο Αχμέτ είναι ένας οικογενειάρχης ο οποίος προσπαθεί να βρει καταφύγιο στην Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν οι ηλικιωμένοι γονείς του Αχμέντα ένας από αυτούς τους φυλακίστηκε για τρία χρόνια. Παρακολούθησα τις λεπτομέρειες στην ε, δίκη του Αχμέτ και η Άμνηστη κατέβαλε κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποφυλακιστεί και να συναντήσει και πάλι την οικογένειά του. Ο Άχμετ δεν είναι τρομοκράτης, αλλά αυτό είναι μια τακτική της κυβέρνησης να να ονομάζει τους ανθρώπους αυτούς ε, τρομοκράτες και να τους ε, συνδέει με εξτρεμιστικές ε, οργανώσεις που επιτίθενται οργανωμένα στη χώρα. Πάρα πολύ ε, συχνά υπάρχει προκατάληψη κατά των μουσουλμάνων και των Αράβων. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να, το, να μας απασχολήσει η χρήση ενός μεγάφωνου και η ρήψη ε, ε, λίθων δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα τόσο σοβαρό αδίκημα. Τα μέλη του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυης ε, την δίκη του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει τις έρευνές της, γιατί εδώ έχουμε μια σαφή παραβίαση. Την κυβέρνηση δεν την απασχολούν μόνο οι μετανάστες, αλλά και οι ίδιοι οι Ούγγροι. Υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις, οι οποίες δεν ε, ε, εφαρμόζονται. Θα πρέπει να δοθούν περισσότερες εξουσίες ε, στον εκτελεστικό κλάδο. Ε, για παράδειγμα, θα πρέπει να μας απασχολήσει το δικαίωμα μετακίνησης και το δικαίωμα έκφρασης στην Ουγγαρία. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να πάρει μέτρα για 15 μέρες, κατεξαίρεση μέτρα, να αναπτύξει το στρατό και να επιτρέψει την χρήση πυροβόλων όπλων. θα μπορούσε να εφαρμόσει ειδικά μέτρα προκειμένου να αποφύγει τρομοκρατικές δράσεις. Νομίζω ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τέτοιες περιπτώσεις υιοθέτηση ακραίων μέτρων. Διάφορες ομάδες πιστεύουν ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει εντελώς αυθαίρετα τα μέτρα αυτά. Κυρίες και κύριοι, το μήνυμα που θα ήθελα να σας στείλω σήμερα είναι το εξής. Αυτό που θέλουμε ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να λάβει υπόψη της και άλλες δράσεις, ενδεχομένως μία επίσκεψη στην Ουγγαρία. Η Ουγγαρία θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα, να μην κάνουμε πολύ λίγα πράγματα και πάρα πολύ αργά. Η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί ότι η κατάσταση στην ε, Ουγγαρία είναι σοβαρή και υπάρχει περίπτωση παραβίασης πολλών κανονισμών. Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει μόνο τη δυνατότητα αλλά και το καθήκον να δράσει. Ευχαριστώ. Ο ομιλητής, η Στεφάνια η οποία είναι εκτελεστική διευθύντρια της Ουγγρικής Ένωσης Πολιτικών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω στην ακρόαση αυτή. Θα ήθελα να εστιάσω στην κατάσταση της ελευθερίας της έκφρασης και ενημέρωσης στην Ουγγαρία. Η ελευθερία ενημέρωσης και έκφρασης είναι μέρος του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να γίνεται σεβαστή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μιλήσω για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ουγγαρία. Μπορούμε να δούμε μια τάση που καθορίζει τον πλουραλισμό, την τάση της αναδιαμόρφωσης της αγοράς των μέσων και της αναδιανομής των πόρων. Ο στόχος είναι κυρίως οι επιχειρήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Χαρακτηριστικό Το υποστηρίζει και το think tank των Media Mertak. Μπορεί να υποθεί πως η κατάσταση στην Ευρώπη το 2014 υπόθηκε πως πολύ λίγα μέσα εταίροι μπορούν να παρατηρηθούν μεμονωμένα. Πολλοί ελέγχονται, κατευθύνονται από επιχειρηματίες με καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Το 2015 μεταξύ άλλων είχαμε την περίπτωση του TV2 ενός τηλεοπτικού καναλιού που αγοράστηκε από ένα στέλεχο της κυβέρνησης το 2015 αγοράστηκε επίσης από έναν επιχειρηματία που είχε καλέσει επαφέ με την κυβέρνηση ένας τηλεοπτικός σταθμός το 2016 μια ανεξάρτητη εφημερίδα έκλεισε ξαφνικά οι εργαζόμενοι απολύθηκαν και τα αρχεία καταστράφηκαν. Ένα δικαστήριο το χαρτηρίσα παράνομα εκ των υστέρων, αλλά η εφημερίδα ήδη είχε διακόψει την κυκλοφορία της. Όλο αυτό εξηγήθηκε με οικονομικούς λόγους, αν και η Media World πούλησε τα μερίδια της κατά 100% και αυτό βάσει στενών επαφών με την κυβέρνηση. Και άλλα έντυπα μέσα σχετίζονται με επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται στην... με σχέση στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να υποδείξουμε και πάλι τις διατάξεις που υπάρχουν, επίσης για την επιχορήγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βλέπουμε ότι γίνεται μια ανομοιόμορφη κατανομή διαφημιστικών μέτρων στην Ουγγαρία. Οι τάσεις αυτές συμβαδίζουν με περιορισμούς Πολλοί δημοσιογράφοι, παραδείγματο χάρη, δεν μπορούν να πάνε στους καταβλισμού προσφύγων. Κατά την προσφυγική κρίση το 2015, μια σειρά δημοσιογράφων και ολόκληρα όργανα του τύπου δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στους χώρους αυτούς. Τους επιτράπει μόνο η πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους, αν και κάποιες από τι απαγορεύσει άρθηκαν και πάλι. Το δεύτερο που θα ήθελα να θίξω σχετίζεται με την κατάσταση των ενεργών πολιτών στην Ουγγαρία, οι οποίοι δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάποια στοιχεία ή σε εκθέσεις δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως σε σχέση με κριτική. Πολλές φορές οι πολίτες αυτοί δέχονται αγωγές, χάνουν τις θέσεις τους ή κατηγορούνται για συκοφάντηση. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται μια αποσιώπηση της αθέμητης κριτικής με αυτόν τον τρόπο πολλοί άνθρωποι πλέον δεν εκφράζονται με κριτικό τρόπο, ιδίω εάν θεωρούν πως αντιμετωπίζουν κίνδυνο καταβολής εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ως αποζημίωση. Ο εντεταλμένος περί ανθρώπινων δικαιωμάτων είπε μεταξύ άλλων πως υπάρχουν πολλές δυσκολίες στον τομέα αυτό Ο νόμος έκανε δυνατή την απόρριψη αιτημάτων πρόσβασης σε πληροφορίες. Είναι ίσως δυνατόν να γίνονται καταβολές χρημάτων όχι μόνο για την αποστολή αιτήσεων. Ανώνυμες αιτήσεις δεν είναι πλέον δυνατές. Το 2016 συνεχίστηκε η κατάσταση αυτή όσον αφορά τις πολιτικές ελευθερίες είχαμε κρατικές επιχειρήσεις και την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας. Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για ανεξάρτητα όργανα να εργαστούν. Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ το 2016 επισκέφθηκε τη χώρα μου. Σε τρεις μέρες θα δημοσιευτούν οι συστάσεις του. Υπέδειξε μία σειρά δυσκολιών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουγγαρία και υποδεικνύει πως οι συνθήκες εργασίας για ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι οι καλύτερες. Το 2013 άρχισαν τα πρώτα προβλήματα, το 2016 φτάσαμε μια νέα κλίμακα όταν ο αντιπρόεδρος του Φέντες και άλλα όργανα του Κοινοβουλίου είπαν σε μια συνέντευξη πως προτρέπουν τις Εθνικές Υπηρεσίες Ασφάλειας και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας να εξετάσουν εκ του σύνεγγυς οργανώσεις που συνεργάζονται με το δίκτυο Σόρος. 22 τέτοιες οργανώσεις ταυτοποιήθηκαν και υπόθηκε πως οι οργανώσεις αυτές παραβαίνουν ουγγρικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν δημοσιεύτηκαν περαιτέρω εκθέσεις αλλά θα πρέπει να υποθεί πως διαπιστώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πως τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουγγαρία δεν γίνονται σεβαστά. Επίσης υποδείχθηκε από διάφορους ανθρώπους πως τα δικαιώματά τους δεν προστατεύονται εάν δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μηχανισμοί ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση. Επίσης υπήρξε στιγματοποίηση οργανώσεων πολιτών στο Κοινοβούλιο για το εαρινό πρόγραμμα το οποίο προβλέπει μια τροποποίηση μιας νομοθεσίας σχετικά με οργανώσεις οι οποίες πρέπει να καταβάλουν συγκεκριμένα στοιχεία για το εισόδημά τους και βάσει διατάξεων από το 2015 πρέπει να θεωρούμε δεδομένο πως η ρύθμιση μέσω ΜΚΟ και οι δυνατότητες παροχής πληροφοριών όσον αφορά το εισόδημα ΜΚΟ, πως αυτές οι διατάξεις πρόκειται να αυστηροποιηθούν. Αύριο θα γίνει μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά, αν και το θέμα είναι ακόμα η δήλωση εισοδήματο. Έω τώρα δεν έχει δημοσιευτεί ένα σχέδιο νόμου. Υπάρχουν όλο ένα και, και και καινούριε ιδέε από κάθε δυνατή κυβερ... κατεύθυνση τη κυβέρνηση με τον στόχο τη βελτίωση τη διαφάνεια των ΜΚΟ. Αφενός προτείνεται η παροχή πληροφοριών οι οποίες πρέπει να παρέχονται ήδη και οι προτάσει αυτές προέρχονται από υψηλό βαθμό στελέχη της κυβέρνηση και από υπουργού. Το θέμα αυτό τέθηκε και από τον Πρωθυπουργό κατά την ομιλία του προς το Έθνος υπάρχουν τρία σημεία κριτικής, πως γίνεται κατεύθυνση από το εξωτερικό, πως μέτρα γίνονται χωρίς κατάλληλη εντολή και ότι χρειάζονται μέτρα για τους χρηματοδότε. Παρότι η οικονομική μας έκθεση είναι δημόσια και περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτές οι οργανώσεις σχετίζονται συχνά με, με, με μια επιρροή στην προσφυγική κρίση. Η πρόθεση της διαφάνειας δεν πρέπει να οδηγήσει σε αυτό, καθώς αυτές οι προτάσεις έχουν ως στόχο τον στιγματισμό ή και την κατάργηση των οργανώσεων αυτών. Στις αρχές Ιανουαρίου ο αντιπρόεδρος της, του κυβερνητικού κόμματος υπέδειξε πως οι οργανώσεις αυτές που έχουν σχέση με το δίκτυο σώρος πρέπει να πεταχτούν έξω από τη χώρα. Η ρητορική αυτή και η τακτική μας είναι γνωστή από το Ισραήλ και τη Ρωσία και ο ειδικό εισηγητής υποδεικνύει επίσης στη μεγάλη ανησυχία που επικρατεί όσον αφορά τη συνεχιζόμενη το συνεχιζόμενο στιγματισμό ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όσον αφορά την επιθετική ρητορική εκπροσώπων της κυβέρνησης σε σχέση με τις οργανώσεις αυτές. Η εκστρατεία εκφοβισμού είναι προβληματική, ιδίως υπό το πρίσμα της ελευθερίας της έκφρασης, που είναι μόνο ένα στοιχείο του προβλήματος αλλά υπάρχει και το στοιχείο του εξωτερικού, δηλαδή της χρηματοδότησης από το εξωτερικό και πώς ορίζεται αυτή, έχει επιπτώσεις για την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, που είναι μια θεμελιώδης ελευθερία. Την περασμένη εβδομάδα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι το κυβερνητικό κόμμα και άλλες ομάδες έχει στοχεύει σε μια ολόκληρη σειρά οργανώσεων και γι' αυτό προσπαθεί να γίνει μια απογραφή με ένα μητρό μίκιο που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό. Ο τελευταίος ομιλητής, η κυρία Μάρτα Παρντάβη, που είναι συμπρόεδρος της ε, Επιτροπής του Ελσίνκη της Ουγγαρίας. Thank Πρόεδρε, κύριε, κύριοι Ευρωβουλευτές, είμαι, είναι τιμή μου να είμαι εδώ και να σας μιλάω. Είμαι συμπρόεδρος της Επιτροπής Ελσίνκη, ε, που είναι μία ΜΚΟ της Βουδαπέστης. Ε, ασχολούμαστε με την προστασία των ε, προσφύγων, την ποινική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου ε, θέματα της αρμοδιότητάς σας. Θα ήθελα να συμπληρώσω τις δηλώσεις της ε, συναδέλφου και να μιλήσω για τα, ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα αυτή τη στιγμή στην Ουγγαρία προστασία των προσφύγων. Τα κράτη φυσικά θα πρέπει να προστατεύσουν τα σύνορά τους, έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη, αλλά έχουν την υποχρέωση να ε, προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων των σύνορων. Ε, θα πρέπει να ε, αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με ανθρώπινο τρόπο, ε, να τους δείχνουν σεβασμό και να σέβονται το δικαίωμά τους να ζητήσουν άσυλο, εξασφαλίζοντάς τους αποτελεσματική διαδικασία ασύλου. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη γίνεται μια συνεχή μάχη για να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο των συνόρων και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αναμφιβόλως είναι πολύ δύσκολο αυτό το έργο. Όμως, ε, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση στην Ουγγαρία, η αναζήτηση αυτή τη ισορροπία και η προσπάθεια για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμό του ενωσιακού δικαίου έχουν εγκαταληφθεί εντελώ από το καλοκαίρι του 2015. Ε, από τον Αύγουστο του 2015 η Ουγγρική κυβέρνηση ε, έλαβε μία σειρά από δραστικά φυσικών και νομικών μέτρων που ουσιαστικά διέλυσαν το σύστημα προστασίας των προσφύγων στην Ουγγαρία. Ο συνδυασμός, ε, η συνδυαστική επίπτωση ήταν αυτά τα μέτρα να αποτρέψουν ε, τους ανθρώπους που θέλουν ε, διεθνή προστασία από το να αναζητήσουν την προστασία αυτή στην Ουγγαρία. Φυσικά όλοι γνωρίζετε τα μέτρα που λήφθησαν. Πρώτον, μιλάμε για μέτρα τα οποία απορρίπτουν, που οδηγούν στην απόρριψη όλων των ανθρώπων που μπήκαν στην Ουγγαρία από την Σερβία ή τα νότια σύνορα, θεωρώντας ότι είναι μη παραδεκτές οι αιτήσει ε, λόγω της αρχής της τρίτης χώρας. Γιατί η κυβέρνηση υπό τη Σερβία είναι ασφαλή σε τρίτη χώρα και επομένω ε, δεν γίνεται καμία προσπάθεια να αναζητήσουν γιατί οι Σύριοι, οι η κυβερνηση απο οι Αφγανοί και άλλοι ε, φεύγουν οι αυγανοι και αλλοι φευγουν απο τις χώρες τους. Ε, νέες και άδικες διαδικασίες έχουν εισαχθεί ε, και το αποτέλεσμα είναι οι πραγματικοί πρόσφυγες να μην έχουν πρόσβαση σε πραγματικές ε, διαδικασίες ασύλου και στη δυνατότητα εξασφάλισης προστασίας. Τα σύνορα σφραγίστηκαν ε, με σειρματοπλέγματα και οι μετανάστε οι οποίοι έχουν περάσει από αυτό το σειρματόπλεγμα τους αποδίδονται ποινικέ κατηγορίες με ταχύρυθμες ποινικέ διαδικασίες χωρίς εγγύηση των δικαιωμάτων τους. Επίσης δεν υπάρχουν ε, ε, επαρκείς ε, συνθήκες υποδοχής. Πολλά στρατόπεδα, μεγάλα ειδικά έχουν κλείσει και η κουρική κυβέρνηση έχει καταφύγει τώρα στο να δίνει έμφαση στην, στην προσωρινή εγκατάσταση, παραδείγματο χάρη αντίσκηνα κτλ., που δεν είναι επαρκή προστασία των ανθρώπων ε, κατά διάρκεια του χειμώνα ή ε, μέσα σε κοντέινερ. Ε, επίσης, Επίση, έχει ανοίξει ένα μικρό άνοιγμα στο σειρματόπλεγμα, στα νότια σύνορα. Ε, ε, είναι μια διαδικασία υποτίθεται διαχείριση τη εισόδου. Όμως το Γραφείο Μετανάστευσης της Ουγγαρίας μόνο, ε, αφήνει μόνο 25 άτομα την, τη εβδομάδα να ζητάνε, να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Ε, Σχεδόν είχε σφραγίσει την πρόσβαση στη χώρα. Το 2016 η κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει νέα νομικά και πρακτικά μέτρα για να αποτρέψει περαιτέρω το, τη ροή των μεταναστών και προσφύγων, αρνώντα την πρόσβαση στην προστασία για του πρόσφυγε. Και από τον Ιούλιο η αστυνομία υποχρεούται να συνοδεύει προς τα πίσω, ε, προς το εξωτερικό στα εξωτερικά σύνορα τους ε, μετανάστες που τους έχουν, αντιληφθεί ε, σε μια περίμετρο ενός χιλιόμετρου γύρω από το σειρματόπλευμα. Ε, στέλνονται δηλαδή προς τη Σερβία οι μετανάστευση και επομένως δεν μπορούν να αναζητήσουν τα άτομα διεθνή προστασία. Αυτά τα άτομα ε, ουσιαστικά βρίσκονται μπλοκαρισμένοι στην Σερβία σε απάνθρωπες ε, συνθήκες γιατί το σύστημα ασύλου της Σερβίας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή ε, τη ροή ας πούμε, τις 7.000 ανθρώπους που θέλουν να, ε, καταφύγιος. 19.000 επίσης ε, άτομα ε, εκδιώχθηκαν προς την ε, Σερβία. Δεν τους καταχώρησε κανένας ατομικά, δεν, τους, δεν υπήρξε καμία απόφαση εξατομικευμένη για την επιστροφή τους, δεν υπάρχει καμία νομική διαδικασία και ένδικα μέτρα ε, ως τμήμα της προσπάθειας αυτής να τους σπρώξουν προς τα πίσω. Φυσικά υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Όταν χιλιάδες λαθρομετανάστες δεν ελέγχονται ή τα δεδομένα τους δεν ελέγχονται με βάση τα όσα είναι καταχωρημένα σε ε, βάσεις δεδομένων. Ε, υποτίθεται ότι ε, χρησιμοποιούνται μόνο οι ειδικέ διαδικασίε που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με καταχρηστικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφύγει εναντίον τη Ουγγαρία, μια διαδικασία που συνεχίζεται. Από την άνοιξη του 2016, τιμή ε, εξακολουθούν να λαμβάνουν ανισχυτικές εκθέσεις για σοβαρές καταχρήσεις ε, και παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά μεταναστών και τουν τον άσυλο. Ε, η Υπηρεσία Προσφύγων του ΟΗΕ, ε, η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν εκφράσει επίση σοβαρέ ανησυχίε για τι καταχρηστικέ αυτέ πρακτικέ και η Frontex επίση παρακολουθεί την κατάσταση. Όμω, οι Ουγγρικέ Αρχέ Σήμερα, ε, μέχρι σήμερα δεν έχουν δείξει διάθεση να κάνουν ε, ουσιαστικές και ενδελεχείς έρευνες για, σε αυτά τα, τα patterns, αυτά τα μοντέλα κατάχρησης των ε, διαδικασιών. Επίσης, ε, βλέπετε αυτές, ε, αυτά τα έγγραφα, ε, τα οποία κυκλοφορούν στην Ανατολική Ευρώπη. Ένα νομοσχέδιο προτείνεται από την κυβέρνηση και βρίσκεται ενώπιον του Κοινοβουλίου για να υιοθετηθεί στην αιρνή Σύνοδο, που θα επιτρέπει στις αρχές αυτόματα να κρατούν οποιονδήποτε ετούντα άσυλο, περνάει από τα σύνορα και να ε, οδηγήσουν τους μετανάστες προς τα πίσω, ε, που θέλουν, άτομα τα οποία θέλουν να ζητήσουν άσυλο, αλλά δεν έχουν νόμο καθεστώς ε, στη χώρα και θα τους επιστραφ, επιστρέψουν στη Σερβία. Οπουδήποτε και αν τους βρουν στην, στην Ουγγαρία, ανεξάρτητα από το σημείο εισόδου τους. Αυτές οι διατάξεις θα ισχύσουν όσο υπάρχει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη μετανάστευση που υπάρχει από το Σεπτέμβριο του 2015. Και ε, έχει επεκταθεί αυτή η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Εάν εγκριθεί το νομοσχέδιο ε, και γίνει νόμος, οι αρχές θα μπορούν να κρατούν όλους τους ενήλικους τούντες άσυλο που ε, κρατούνται στην επικράτεια, ακόμα και γυναίκες με παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι πάνω από τα 14 χρόνια. Επίσης, δεν θα υπάρχουν ασφαλείς ζώνες ε, και επίσης δεν θα υπάρχουν ένδικα μέτρα για να μπορούν να αμφισβητήσουν αυτά τα μέτρα. Και αν ναι, οι αρχές ε, θα μπορούν ε, με συνοπτικές διαδικασίες να επιστρέφουν τους μετανάστες και τους ετούντες άσυλο ως, όταν μένουν χωρίς άδεια στην Ουγγαρία προς τα σερβικά σύνορα. Και αν εγκριθεί για να μπορέσει να ζητήσει προστασία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ε, τι ζώνε διέλευση του συστήματο ασύλου, εάν σου πούν OK για την ε, είσοδο. Ε, Όμω, ε, όπω σα είπα, μόνο 25 άτομα τη βδομάδα ε, μπορούν να ε, εισέλθουν στη χώρα. Επομένω, δεν ξέρω πόσα άτομα θα μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτή την εγκεκριμένη είσοδο στην χώρα. Οι, χώρες, οι ζώνες διέλευση, όπως είπε η κυβέρνηση, θα έχουν και στέγαση Μιλάμε για 200-300 άτομα. Άτομα από σημερινά κέντρα υποδοχής που είτε είναι ανοιχτά είτε κλειστά θα μεταβούν σε αυτά τα νέα κέντρα. Ε, θα υπάρχουν εξαιρετικές ε, διαδικασίες συνόρων για όλη τη χώρα και θα επιτρέπεται η αυτόματη κράτηση ε, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της ε, αίτησης ασύλου και η, τρίτη, η τρίτων χωρών χωρίς νόμιμη, νόμιμο καθεστώς ε, μπορούν να επωφεληθούν μόνο από κάποια εξαιρετικά μέτρα ε, και αυτή η κράτηση θα, αφορού, θα αφορά όλους τους ανήλικους ε, και τους ασυνόδευτους ανήλικους πάνω από τα 14. Ε, αυτό όμως ε, ουσιαστικά παραβαίνει ουσιαστικά το δίκαιο για τα δικαιώματα των παιδιών και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του παιδιού. Ε, πιστεύουμε ότι ο ε, οι συνδυασμένες επιπτώσεις αυτής της νομοθεσίας ε, θα αναγκάσουν τα ε, άλλα κρατημέλη να μην επιστρέψουν στην Ουγγαρία κανέναν άλλον τούντα άσυλο με βάση τον ε, τον κανονισμό των δουβλίνων και επομένως θα υποσκαφθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Το Human Rights Watch ζητάμε από τον Επίτροπο Αβραμόπουλο σήμερα να εξετάσει την, το νομοσχέδιο αυτό και να λάβει ταχύτατα δράση, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η Ουγγαρία θα σεβαστεί ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο ασύλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ομιλητές. Λόγω της ευαισθησίας και της ε, σημασίας του θέματος θα ήθελα να δώσω σε όλους ε, την ευκαιρία να μιλήσουν. Βεβαίως δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τον κανονισμό μας τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΕ, αλλά προκειμένου να μιλήσετε μπορείτε να πάρετε το λόγο μόνο για 1,5 λεπτό. Αυτό το λέω γιατί θα πρέπει να υπάρξει επαρκής χρόνος, ε, δηλαδή τουλάχιστον 30 λεπτά, από τους συναδέλφους από την κοινωνία των πολιτών. Όλοι οι συντονιστές, ε, όλες οι ομάδες θα πρέπει να εκπροσωπηθούν. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο σε κάποιον από μία πολιτική ομάδα. Έχω 15-16 ομιλητές εγγεγραμμένους. Ε, όλοι οι παριστάμενοι υπάρχουν στον κατάλογο. Κύριε, κύριε Βεζιά, θέλετε να πάρετε το λόγο, ναι ή όχι. Θέλετε. Ωραία, παρακαλώ, είστε στον κατάλογο. Ωραία, ξεκινάμε με το ΕΛΚ, με Τσουρενάκη. Όχι. Πέστε μου σας παρακαλώ για να σας καταλάβω. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι εσείς. Δεν είστε στην ε, Επιτροπή Λίμπε. Α, κανένας άλλος. Ωραία. Ε, σας ζητώ συγγνώμη. Εσείς, εσείς πρώτος κυρία, Παρακαλώ, μιλάτε εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Η ερωτήση μου απευθύνεται στον Υπουργό Δικαιοσύνη και θα ήθελα να γνωρίζω τι μέτρα έχει λάβει η Ουγγρική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις ε, φυλακές και τον μεγάλο αριθμό τροφίμων. Θα ήθελα να ε, γνωρίζω όταν ε, μετρώνται ε, συγκεκριμένε παράμετροι από, για τη δικαιοσύνη, τι αποτέλεσμα έχουμε. Μήπως θα μπορούσατε να επεκταθείτε περισσότερο σε ό,τι αφορά τα συνταγματικά δικαστήρια και τις εξουσίες που έχουν ως πρώην δικαστής, θα μπορούσατε να μας τα δώσετε, θα τα καταλάβουμε ενδελεχέστερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σύντομοι, κυρία Σίπελα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, καθώς μιλούσαν οι ομιλητές, κοίταξα περαιτέρω το θέμα, γιατί με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα για το κράτος δικαίου. Κοιτάζοντας, βρήκα το κέντρο των αθενιδιωτών δικαιωμάτων, έγινε το 13 ενώ βρέθηκαν δύο ονόματα, το δικό σας και ενό άλλου. Και όλα τα άρθρα στη σελίδα έφεραν την υπογραφή του Κέντρου των Θεμελιδιών Δικαιωμάτων. Υπάρχει μια έλλειψη διαφάνειας εδώ. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε πόσοι εργάζονται σε αυτό το κέντρο και πόσοι ε, υπογράφουν αυτό το άρθρο. Με εξπέκλησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο κ. Στροσάνη μίλησε, είπε ότι όλες οι κυβερνήσεις ήταν εκλεγμένες. Κανένας δεν είπε το αντίθετο. Βεβαίως εκλεγμένες, αλλά αν κανείς είναι εκλεγμένος και ανεξάρτητα από τις πλειοψηφίες, θα πρέπει να σέβεται τις διαφορετικές απόψεις, τις διαφορετικές ομάδες, τις διαφορετικές θέσεις θέσεις των ΜΚΟ και των πολιτών. Σε μια δημοκρατία θα πρέπει να έχετε τη βεβαιότητα ότι εκπροσωπούνται και εισακούνται ως σε διαφορετικές απόψεις. Ελευθερία των ΜΜΕ, ελευθερία της έκφρασης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ακόμα πιο σημαντικό σε μια δημοκρατία είναι τα ΜΜΕ να έχουν τη δυνατότητα να επικρίνουν το τελευταίο σημείο για τη διαδικασία ασύλου. Είπατε ότι πολλοί πρόσφυγε θα επιθυμούσαν να έρθουν στην Ευρώπη από ότι να παρεμείνουν σε άλλε ασφαλείς χώρες. Συνειδητοποιείτε ότι οι περισσότεροι πρόσφυγε δεν πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε προστατεύσετε τα σύνορα. Θαυμάσια. Παράλληλα όμω δεν επιτρέπετε στου ανθρώπου αυτού που κρούν τη θύρα και λένε γονάγια από βοήθεια ε, να μπουν μέσα και να τους προσφέρετε καταφύγιο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη συνθήκη της Γενέμης. Το μήνυμα που στέλνετε είναι πηγαίνετε όπου θέλετε, αλλά μην έρχεστε στην Ευρώπη και αν μη τι άλλο μην έρχεστε στην Ουγγαρία. Αυτό έχει σχέση με τη σύμβαση Γενέμης. Δύο λεπτά ακόμα. Πραγματικά πιστεύω ότι το νέο αυτό δίκαιο που ε, θα, θα, θα, εφαρμοστεί, που οδηγεί στη ε, φυλακή τους ε, του άσυλο. Κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μ' ακούτε. Μου έκαναν εντύπωση κάποια από τα λεγόμενα του κύριου Γκάρντος. Αναφέρατε διάφορες ε, διοικητικές διαδικασίες, αλλά κυρίως αναφέρατε απόψεις, γνώμες, δηλώσεις. Όταν ακούτε όταν ακούτε γνώμες από ανθρώπους στο δρόμο, ακόμα και αν αντίθετες με τα όσα ε, λέει η νομοθεσία μας, θα πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους. Ε, επίσης, Θεωρείτε ότι ο κομμουνισμός στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες ήταν ένα σύστημα καταπίεσης και κοινωνικών διακρίσεων που κατέστησε ολόκληρες ομάδες κοινωνικές ε, ε, πολίτες δεύτερης κατηγορίας που τους θεώρησε εχθρούς ή προδότες κτλ. Συμφωνείτε επίσης ότι οι διάφοροι κύκλοι που συνεργάστηκαν με το κομμουνιστικό καθεστώς στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες αφότου κατέρευσε το κομμουνιστικό σύστημα και επανήλθε η δημοκρατία, αυτοί οι κύκλοι χρησιμοποίησαν ακόμα και μετά την ε, ισχύ τους, την εξουσία τους, ε, τα λεφτά τους, να, για να μπλοκάρουν διάφορες αλλαγές, για να, για να μπλοκάρουν ακόμα την χειραφέτηση και την απελευθέρωση διαφόρων κοινωνικών ομάδων, ε, οι οποίες ήταν θύματα του κομμουνιστικού καθεστώτος. Επίσης, συμφωνείτε, όλα αυτά τα είπε η Διεθνής Αμνηστία, έτσι. Συμφωνείτε επίσης ότι κάθε κυβέρνηση που θέλει να προστατεύσει το κοινό καλό θα πρέπει να προστατεύει και τις ομάδες που στο παρελθόν έπεσαν θύματα διακρίσεων. Και ακόμα μία ερώτηση. Γιατί δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά. Τι έχετε να πείτε για την έκτρωση. Πιστεύετε ότι είναι δολοφονία ε, του παιδιού, θεωρείτε ότι είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτό. Ο πρόεδρος εκτός μικροφώνου για απάντηση. Ε, θα ξεκινήσουμε την Πυργίτε. Ε, εγώ δεν μιλάω για το περιεχόμενο, μιλάω για το χρόνο, έτσι. αν όλοι κάνουν δηλώσεις, αν πούνε οτιδήποτε, αν κάνουν ερωτήσεις κτλ. θα είναι δυόμιση λεφτά, τίποτα παραπάνω, έτσι. Γιατί έχουμε μέχρι τις 5 και θέλω να δώσω χρόνο για απαντήσεις. Εάν θέλετε να συνεχίσουμε έτσι, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλιώς θα σας παρακαλώ. Αν θέλετε πραγματικά να συνεχίσουμε όμως όπως πρέπει, μέχρι 1,5 λεπτό. Ε, και θα χρησιμοποιήσω το σφυράκι. Όλοι θα πρέπει να σεβαστούν το, το 1,5 λεπτό αυτό. Ε, την ΚΟΕ, η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε ένα νέο συντονιστή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ δώστε στο Άλτε το λόγο όταν έρθει η σειρά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, υπάρχει ένταση στην αίθουσα και έγινε ένα λάθος. Νάταλη, συγχαρητήρια που έγινε η νέα συντρονίστρια του Άλτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ. Και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα συγχαρητηριά σας. Το σύντομο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου θα είχα να διατυπώσω πολλές ερωτήσεις, ήδη όμως οι συνάδελφοι έθιξαν την ουσία του προβλήματος. Θα ήθελα να πω ότι οθετήσαμε μια νέα οδηγία την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο που αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας προκειμένου να εναρμονίσουμε το ποινικό πλαίσιο σε επίπεδο ευρωπαϊκό μεταξύ όλων των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατία μετά από αυτό που ανέφερε ανέφερε ο εκπρόσωπος του, της Amnesty International μιλώντας για τον Αχμέντά, το ο οποίος θεωρεί το ύποπτος για τρομοκρατικές ενέργειες από τις αρχές της Ουγγαρίας, απλά και μόνο γιατί κρατούσε ένα μεγάφωνο. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψη των Ουγγρικών αρχών και κατά πόσο θα μπορούσαν να μου απαντήσουν ως πρώτη συμβατότητα των αποφάσεων που ελήφθησαν με ευρείας ε, έγκριση ως προς την ανάγκη για αναλογικότητα και ως προς την εγγύηση που παρέχεται για το σεβασμό των ε, ε, ανθρωπίων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να έχουμε και το ένα και το άλλο. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε στην Ευρώπη και να μην εφαρμόζουμε πράγματα που αφορούν εμάς όλους τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ και πάλι. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και συγγνώμη για το λάθος. Η κυρία Πισπινέλη έχει το λόγο τώρα. Πρόεδρε, σας ζητάω να δώσετε το λόγο στην κυρία Βερζιά, γιατί είναι σκιώδη συγγήτρια και εγώ θα μιλήσω μετά από εκείνη. Ωραία, κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το μπέρδεμα. Και ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένη. Εξού και το πρόβλημα. Θα ήθελα να επιμείνω πάρα πολύ στο θέμα με το, ε, ε, που αφορά τους ε, μετανάστες, πώς αντιμετωπίζονται στην Ουγγαρία. Και να μιλήσω για αυτή την δίκη, για μια δίκη που έγινε στην Ουγγαρία. συνολικά τα άτομα τα οποία δικάστηκαν σε αυτή τη δίκη ήταν Σύριοι, δύο από αυτούς είναι άτομα με ειδικέ ανάγκες, ε, ε, ε, έμειναν ανάπηροι ε, μετά στον πόλεμο και η ε, κατάσταση τους ήταν τραγική. Ο Χαμέν Άσου και ο Χαμέν Χα πήραν τις πιο βαριές ποινέ. και οι ποινέ αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι χρησιμοποίησαν μεγάφωνα. Με αυτόν τον τρόπο τους ε, τους κατηγόρησαν για τρομοκρατία. Είναι εντυπωσιακό ο λόγος για, για, τον οποίο κατηγορήθηκαν για τρομοκρατία. Ο Χάμετ Χάς ε, έπεσε θύμα διακρίσεων κατά τη διάρκεια της δίκης του και κατηγορήθηκε για τρομοκρατία, κυρίως γιατί ήταν μουσουλμάνος και όλοι ξέρουμε ότι μερικοί δεν δέχονται τους μουσουλ, μουσουλμάνους. Ε, υπερασπίζονται υποτίθεται την ε, ελευθερία, τη θρησκευτική ελευθερία, αλλά θρησκευτική ελευθερία δύο ταχυτήτων. Επίση, η Ουγγρική κυβέρνηση θέλει να μα πει γιατί σε αυτά τα πλαίσια αυτή τη δίκη ε, δεν ε, δέχτηκε την διαμεσολάβηση του ΟΗΕ και γιατί οι πήκοοι τρίτων χωρών ε, δεν αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο χώρο. Κυρίω ε, να μου πείτε αν αυτοί που έρχονται από την Ανατολική Ουγγαρία ε, και αυτοί που έρχονται από την νότια Ουγγαρία, δηλαδή έχουν περάσει μέσα από τη Σερβία, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Όχι, αν δείτε τα νούμερα, όλων αυτών που φτάνουν στην Ουγγρική επικράτεια, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Ε, ευχαριστώ Α, για τους πράσινους, κυρία Σαρτζεντίνη. Sorry, Chair. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η ερώτησή μου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Ουγγαρίας από ό,τι κατάλαβα έχετε ένα μέτ μια δέσμη μέτρων για τη διαχείριση των σύνορων και των προσφύγων, για το οποίο θα συζητήσετε γύρω στις 7 Μαρτίου, ή ίσως και πιο πριν. Στη δέσμη μέτρων αυτήν, από ό,τι κατάλαβα, περιέχεται η διαδικασία για την αίτηση ασύλου, είναι μια διαδικασία στα σύνορα, η οποία υπάρχει ήδη, μια συνοριακή διαδικασία καταλαβαίνω σωστά πως η κανονική διαδικασία ασύλου δεν θα λάβει ποτέ πια χώρα στην Ουγγαρία και πως όλα θα γίνουν στα σύνορα. Θα ήθελα να το καταλάβω. Επίσης θα ήθελα να καταλάβω πως προβλέπετε το μέλλον των τροπολοποιών αυτών καθώς αποτελούν σαφή παράβαση του ευρωπαϊκού κεκτημένου ήδη είπατε πως αναμένεται μια απόκληση απόψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όταν την βλέπετε να έρχεται μπορείτε να μας πείτε γιατί το, την αιτιολογία της συγκεκριμένης ατιμαχίας. Και τέλος, Πρόεδρε, ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών σε μια δημοκρατία είναι πολύ σημαντικός. Ήδη κάνετε τις ΜΚΟ να περνούν από μια ολόκληρη διαδικασία διαμόρφωσης και θα ήθελα να καταλάβω κατά πόσον υπάρχουν και άλλα σχέδια μείωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Καλ. Θα ήθελα να θέσω μια σειρά ερωτήσεων και πιστεύω πως όλοι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν τη συζήτησή μας στα ουγγρικά, αν και θα διαπιστώσουμε πως υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που δεν ισχύουν ή ερμηνεύονται λάθος, επειδή ακούγονται πολλές δηλώσεις που δεν έγιναν κατανοητές σωστά από κάποιους εκπροσώπους ΜΚΙΟ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου σε σχέση με αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας εδώ. Υπόθηκε πως υπάρχει μια δικαστική απόφαση η οποία δεν είναι αποδεκτή και πως θέλει να ασκήσει πίεση για την άψη της απόφασης. Ξέρετε, όταν συνελήφθη ο Αχμετ είχε περισσότερα διαβατήρια με θεωρήσεις από τον χώρο του Σέγγεν, είχε ένα διαβατήριο της Κύπρου, είναι κάτοχος πέντε σκαφών στην Κύπρο, οπότε πολλοί διερωτώνται τι έκανε στα αυστροσερβικά σύνορα με πέτρες στα χέρια και με ένα μεγάφωνο. Υπήρξαν και πολλοί τραυματισμοί αστυνομικών. Πέντε τραυματίστηκαν και μπορώ να σας πω πως δεν υπάρχει χώρα στην οποία κάποιος δεν θα καταζικαζόταν ο οποίος άσκησε βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων και θεωρώ πως δεν είναι αποδεκτό η Διεθνής Αμνησία να παίρνει μια τέτοια θέση. Πιστεύω πως ο Αχμέτ δεν είχε κανένα λόγο να βρίσκεται εκεί. Και αν βρέθηκε εκεί, είχε τους δικούς του ιδιαίτερους λόγους. Λέμε για την Ουγγαρία. Θέλω να θέσω μία ερώτηση, μία ερώτηση στον Υπουργό, ή μάλλον τρεις ερωτήσεις και θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις. Υπάρχει πρόβλημα με τους πρόσφυγες στην Ουγγαρία, εμείς θεωρούμε. Αλλά η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους πρόσφυγες. Εν τι αυτή η περιπτώση, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα με τους πρόσφυγες, γιατί κάνετε τροποποίησεις του νόμου, γιατί κλείνετε τους μετανάστες σε κοντέινερ κτλ. Επίσης, Πώς σχολιάζεται το εξής. Ότι αυτές οι αλλαγές θα αφορούν και τους νέους πάνω από την ηλικία των 14 χρονών. Τα οποία, δηλαδή άτομα πάνω από τα 14 χρόνια, δεν θεωρούνται παιδιά και θα δικάζονται και θα υποπίπτουν στις ίδιες διαδικασίες με τους ενηλίκους. Και γιατί εκνευρίζεστε ή ενοχλείστε όταν ε, οι ΜΚΟ εκφράζουν τι απόψει του ή προσπαθούν να επηρεάσουν τα πράγματα. Ακριβώ αυτό δεν είναι δημοκρατία. Ο καθένα να εκφράζεται και εν στοιχεία ε, το εκλογικό σώμα αποφασίζει τι προτιμάει. Γιατί πιστεύετε ότι μόνο οι αιρετοί εκπρόσωποι μπορούν να μιλάνε για την πολιτική και να εκφράζουν γνώμη για την πολιτική στην Ουγγαρία. Κυρία Κατρίκα. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις απευθυνόμενοι στον Υπουργό. Πρώτη ερώτηση. Πράγματι, η κυβέρνηση είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης κομμουνιστικής εποχής, όπως μας έδωσε να καταλάβουμε ο κύριος Γιούρεκ, φαίνεται ότι στην ουγγρική κοινωνία υπάρχουν ε, πάρα πολλά χρώματα και η κομμουνιστική αντιπολίτευση κινείται σε ένα άλλο μέτωπο. Ο Υπουργό είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει διακρίσεις για τις επιχειρήσεις. Πεςτε μου κάτι, ποιες χώρες ε, αποτελούν ε, θύματα διακρίσεων και για ποιο λόγο. Κύριε Γιώζα. Οι συνάδελφοί μου ήδη ανέφεραν τον προβληματισμό τους ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Ουγγαρία. Αυτό βλέπουμε, το βλέπουμε στον εκφοβισμό των ε, ΜΚΟ, ε, το γεγονός ότι συρρυκνώνεται ο αριθμός τους, ε, τη σχέση με τα ΜΜΕ κτλ. Και βεβαίως την κατάσταση ως προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κι άλλες επιπτώσεις. Οι επιπτώσει αφορούν την καταπολέμηση τη διαφορά, σαν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η κοινωνία των πολιτών δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα αποκάλυψη αυτών των θεμάτων και τα ε, ΜΜΕ αποτελούν θύματα τρομοκρατία. Στη χώρα μου πρόσφατα ήταν μία έκθεση για ένα μικρό τρένο που δεν πηγαίνει πουθενά. Στην πατρίδα του, του Πρωθυπουργού Ομπάνα. Ένα τρένο χρηματοδοτείται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ερώτησή μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τι κάνει η Επιτροπή αναρωτιέται τι γίνεται με τα κοινοτικά κονδύλια. Δεν μιλάμε μόνο για διαφθορά στην Ουγγαρία. Ένα από τα θέματα που μας απασχολούν είναι οι φόροι. Οι φόροι όμως είναι κάτι που μπορούσαμε να ορίσουμε μόνο όταν συνεργαζόμαστε, όχι ακολουθώντας την πορεία της Ουγγαρίας. Πιστεύω ότι ότι οι διάφοροι φορείς ανάπτυξης της Ουγγαρίας στέλνουν ένα μήνυμα ότι η Ουγγαρία είναι μια χώρα η οποία διαμεσολαβεί στο ξέπλυμα χρημάτων. Αυτές είναι ερωτήσεις που θέτω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολύ περισσότερο παρά στην Ουγγρική κυβέρνηση. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ να διώξετε από τη χώρα φτωχού και αντιπεράσπιστους ανθρώπους και όχι μερικούς ολιγάρχες που έχουν εγκατασταθεί χωρίς κανένα πρόβλημα στην Ουγγαρία. Δεν είναι η μοναδική χώρα, αλλά όνειδος παραμένει σε κάθε περίπτωση. Ο κύριος Πίστεσεν, παρακαλώ. Για να είμαι ειλικρινής. Για να είμαι ειλικρινής, αυτή η συζήτηση ανήκει στο Ουγγρικό κράτος και θα πρέπει να γίνει εκεί κατά την απόψή μου. Είναι αστείο που κάποια από τα παραδείγματα που ανέφερα μπορούν να βρεθούν σε παρόμοιο βαθμό και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτου ανάγκη λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων εδώ και καιρό και πιστεύω πως αυτή είναι μια συζήτηση που άπτεται των κρατών μελών και αλλού έχει γίνει αναδιανομή των πόρων για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Δανία παραδείγματος χάρη σε άλλες χώρες. Καθώς όμως πολλοί επιμένουν αυτή η συζήτηση να γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντί για το Ουγγρικό Δημοκρατικό κράτος, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό. Το μοντέλο επανοπροθήσεων που αναφέρατε προς την Σερβία, την οποία χαρακτηρίσατε ως ασφαλές τρίτο κράτος. Αυτό δεν είναι πολύ παρόμοιο με αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Ευρωπαϊκή Κλίμακα. Και μπορείτε να αναφερθείτε σύντομα στη συμφωνία που επιτεύχθη με την Τουρκία σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. Καθώς από ό,τι φαίνεται από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καλύτερη στην Τουρκία από ό,τι στη Σερβία. Και για την προσωπική μου άποψη η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία είναι κατά πολύ χειρότερη από τη στην Σερβία, αλλά σας μπορείτε να πείτε κάτι σχετικό. Η κυρία Γουίξτρομ, παρακαλώ, συγγνώμη για το πέδεμα πριν. Ευχαριστώ πολύ. Ρητός, λοιπόν, ακούσαμε από συναδέλφους και από τους καλεσμένους μας από την Ουγγαρία πως υπάρχει η αίσθηση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει επειδή δεν έχουμε αρμοδιότητες στις περιπτώσεις αυτές και πως η Ουγγαρία λίγο πολύ επιλέγεται. Λυπούμε γι' αυτό. Είμαστε μια οικογένεια κρατών μελών και ανθρώπων και πρέπει να αλληλοϊποστηριζόμαστε, επίσης σε δύσκολους καιρούς. Πιστεύω πως το άρθρο 2 βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεών μας και πως οι αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης κτλ. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ανησυχητικό. Είναι η κατάσταση των μεταναστών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, εργαζόμαστε επί της αναθεώρησης του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Είμαι εισηγήτρια για τον κανονισμό του Δουβλίνου. Αυτό θα υπάρχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το από το ποια χώρα θα εξετάσει τα αιτήματα ασύλου και μέχρι τους μηχανισμούς αναδιανομής, στους οποίους θα συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Πώς είναι δυνατόν πως τα μηνύματα που ακούμε από το Συμβούλιο είναι ανησυχητικά. Θα ήθελα να, σα να σας ακούσω, να επισέλθετε λίγο περισσότερο στο θέμα αυτό, έχοντας κατά νου αυτό που είπε κάποιος, πως 85% των εκατομμυρίων προσφύγων στον κόσμο επί του παρόντος βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έρχεται στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε μια κατάσταση στην οποία κάθε κράτος μέλος δεν αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης του. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Ήταν απαραίτητη. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερος της ΜΚΟ για τις μαρτυρίες τους που δείχνουν ότι εδώ και έξι χρόνια χωρίς καμία σοβαρή αντίδραση της ε, Ευρώπης η κυβέρνηση της Ουγγαρίας κάνει έτσι, αυταρχικές παρεμβάσεις ε, που σκοτώνουν τις ελευθερίες. Εγώ δεν θεωρώ ότι το να υπερασπιζόμαστε τον αξιοπρεπή μισθό, ας πούμε, ε, παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και το δίκαιο για την απόσπαση των εργαζομένων. Ε, έχετε επίσης ε, ξενόφοβη ρητορική με σκοπό να αυξήσετε το μίσος και το μίσος εναντίον της Ευρώπης. Ε, αυτή η κατάσταση είναι τρομοκρατική. Ο κύριος Ορμπάν μιλάει ότι θέλει να ε, οδηγεί σε κράτηση τους ανθρώπους που βρίσκονται ε, στην επικράτεια του, της, της Ουγγαρίας. Ε, απευθύνομαι σε εσάς ΜΚΟ. Ε, τι περιμένετε από εμά, τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΜΚΟ. Είδατε, ε, η επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία είναι αντίστοιχη με της Πολωνίας και δυστυχώς η Κομισιόν παρότι έκαν ξεκίνησε μια διαδικασία επί παραβάση κατά της Πολωνίας δεν το έκανε για την Ουγγαρία λόγω τεχνικών λόγων ας πούμε και γιατί ο κύριος Ορμπάν ε, ανήκει στο ΕΛΚΑ. Ε, Όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι αποφασιστική ε, πέρα από τέτοιε διαιρέσει. Θα πρέπει να σέβεται τα θέματα δικαιώματα και ε, να αναγκάζει τις χώρες και πριν και μετά την ε, ένταξή τους να σέβονται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ε, περιμένουμε η Κομισιόν να κάνει το έργο της και θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, που θα ελέγχει την κατάσταση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή μου προς τον, προς τον κύριο Υπουργό είναι αφορά την κατάσταση των γυναικών, τις εκτρώσεις, την Επιτροπή της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των γυναικών και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ποια είναι η κατάσταση σχετικά με αυτό. Κυρία Φιλέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να απευθυνθώ στους εκπροσώπους της αγγουρικής κυβέρνησης και της, θέλω να τους πω, δεν έχει νόημα να, ε, να θυμηθούμε τα θύματα του κομμουνισμού ε, εάν η περάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρείται πολιτική ορθότητα. Αν αυτός ο ορισμός των δικαιωμάτων αυτών θεωρείται ότι είναι στην διακριτική ευχαίρεια του κάθε κράτους μέλους. Η Ένωση όντως δεν έχει το δικό της Δήμο, αλλά αποτελείται με βάση αυτό που λέμε ε, συνταγματικό πατριωτισμό. Δηλαδή, να σεβόμαστε το κράτος δικαίου, το, τη χάτα δικαιωμάτων, τη σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από αυτή την άποψη ε, είμαι ευγνώμων προς το Human Rights Watch και την Επιτροπή του Ελσίγη για την επιστολή που έστειλαν προς τον κύριο Αβραμόπουλο και θέλω να επικεντρωθώ σε κάποια θέματα του νέου νόμου για την προστασία των συνόρων που ελπίζω ε, θα αναθεωρηθεί. αυτό το νομοσχέδιο μιλάει για αυτόματη κράτηση στις χώρες διέλευσης και οφείλεται στο κράτος εκτάκτης ανάγκης, λέει. Ε, υπάρχει εδώ και ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο αυτό το κράτος έκτακτης ανάγκης και τα κριτήρια είναι τελείως θολά. Η κρίση, η μεταναστευτική, δεν είναι μεταναστευτική κρίση, αλλά είναι κρίση της Ευρώπης απέναντι στους ε, μετανάστες. Ένα άλλο ερώτημα που θα ήθελα να κάνω αφορά τις διαδικασίες για την διάθεση που έχετε να πληρώσετε το κόστος της κράτησης στους εκτούντες άσυλο και την αδυναμία να χρησιμοποιήσει κανείς ένδικα μέσα σε περίπτωση που θεωρηθεί είναι παραδεκτή αίτησή του. Ε, θα ήθελα να μου πείτε πώς συμβα... Ε, συνάδει αυτό με το διεθνές δίκαιο. Ο κύριος τέλος. Ένα μέρος της ερώτησής μου αφορούσε την περίπτωση Αχμέτ. Δεν θέλω να σας ε, διορθώσω. Ε, ε, το θέμα της διαφθοράς αφορούσε ένα, το μετρό, όχι ένα μικρό τρένο. Μια, αυτή τη μικρή διόρθωση θέλω να κάνω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ συνάδελφοι για που δείξατε τόσο σημαντικά και ευαίσθητα θέματα. Αρκετές από τις ερωτήσεις σας ε, τις απευθύνατε στον Υπουργό, ο οποίος θα πάρει το λόγο για να απαντήσει. Μερικές παρεμβάσεις αφορούσαν σχόλια και δεν ήταν ερωτήσεις. Θα χρησιμοποιήσω τα 35 αυτά λεπτά όσο γίνεται καλύτερα. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους από τις διάφορες οργανώσεις να πάρουν πρώτα το λόγο, να κάνουν τα σχόλιά τους πάρα πολύ σύντομα και ο υπουργό θα πάρει δεύτερο το λόγο και θα απαντήσει στα ερωτήματα που ετέθησαν. Αυτό είναι και αίτημα των συναδέλφων και όχι μόνο του Υπουργού. Δεν θέλω να πάρετε όλοι το λόγο γιατί ο χρόνος πιέζει. Σας παρακαλώ πολύ αποφασίστε ποιος από εσά θα πάρει το λόγο. Δύο-τρία λεπτά είναι ο μέγιστος χρόνος αγόρευσης. Δύο λεπτά το πολύ ο καθένας, παρακαλώ. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο πρώτος. Παρακαλώ. Κύριε Πεντάβη, Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, για τα σχόλια και για τους προβληματισμούς σας σε ό,τι αφορά τη θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στο θέμα της κράτησης των ετούντων άσυλο. Κατά την άποψή μου είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό θέμα. Όχι μόνο γιατί θα πρέπει να είναι ένα έσχατο μέτρο, αλλά και γιατί θα πρέπει να αξιολογείται η ανάγκη της αναλογικότητας της απόφασης, προκειμένου να υπάρξει κράτηση. Μεταξύ των άλλων, επηρεάζει και ένα μεγάλο αριθμό ετούντων άσυλο στην Ουγγαρία. Η Ουγγαρία ήταν πάρα πολύ γνωστή ότι συχνά κρατούσε τους ετούντες άσυλο, φυλάκιζε τους ετούντες άσυλο. Στις ε, περιοχές ε, διέλευσης δεν έχει ληφθεί μία απόφαση κράτησης. Τα ΜΜΕ στην ε, Ουγγαρία το κατέστησαν σαφές ότι δεν εξετάζεται καν και το ενδεχόμενο της στέρησης ελευθερίας δεν, όλα αυτά δεν εφαρμοζόντουσαν το, τώρα, δεν εφαρμοζονται τώρα και δεν θα εφαρμοστούν και στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη βασανιστήριων εξέτασε βεβαίως αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια της τελευταίας της επίσκεψης στην Ουγγαρία και εκτενώς αναφέρθηκε τις συνθήκες κράτησης στην Ουγγαρία. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σαφές ε, σε όλους ότι αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε, σε μια κράτηση, σε κρατήσεις. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις περιπτώσεις κατά περίσταση και θα πρέπει να ε, βρεθούν διάφορα μέσα. Ε, ένδικα μέσα παροχή νομικής βοήθειας, ε, Τίποτα από αυτά δεν προβλέπεται. Οι αιτούντες άσυλο καλούνται να πληρώσουν για τις ε, δαπάνες της κράτησής τους, εκτός αν υπάρξει μια θετική απόφαση ως προς την ανάγκη παροχής διεθνούς προστασίας. Σας ευχαριστώ πολύ που θα παρακολουθήσετε αυτά τα θέματα σε συνεργασία με την Ουγγρική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Στεφάνη Καπρόνσκια. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες που εκφράζετε. Σε ό,τι αφορά για την, τα ΜΜΕ, υπάρχει ένας κανονισμός για να περιοριστούν τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει η τάση ε, περιστολής του πλουραλισμού ε, και λογοκρισίας. Ορισμένες γνώμες, ε, οι γνώμες που εκφράζονται από κάποιο κοινό, ε, χειραγωγούνται. Αυτό θα πρέπει να μας ε, ε κρούει τον κόδωνα. 87% των δημοσιογράφων ε, πιστεύουν ότι ε, η πολιτική αυτή που ελέγχει τα ΜΜΕ και όχι το αντίθετο. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει για την κοινωνία των πολιτών και την σχετική νομοθεσία, μην ξεχνάμε ότι όταν στυλιτεύουμε τι ΜΚΟ, γιατί εκφράζουν την γνώμη του ε, και ασκούν την ελευθερία, το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης, αμφισβητούμε την ίδια τη φύση της δημοκρατίας. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω περισσότερο για τον προτινόμενο κανονισμό για τα ΜΜΕ και να ακούσω περισσότερα για τον προτινόμενο κανονισμό ε, για την κοινωνία των πολιτών. Καλύτερα, όχι τα, τα ΜΜΕ, την κοινωνία των πολιτών είναι ο κανονισμός. Ο κ. Γκάρντος, τα εγκλήματα επί κομμουνιστικού καθεστώτος συνέβησαν και θα πρέπει να τα διερευνήσει κανείς. Ε, και μου κάνει εντύπωση που το ακούω αυτό από σας κύριε Γιάρκος, γιατί διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, ε, διερεύνησαν το θέμα, αλλά ποτέ δεν καταλήξαμε σε απόφαση. σε ό,τι αφορά την έκτρωση, η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να παίρνουν απόφαση για το σώμα τους και να αποφασίζουν αν θέλουν να συνεχίσουν την εγκυμοσύνη τους ή όχι. Η προστασία του εμβρίου ε, ε, εξασφαλίζεται από την αρχή της δεκαετίας του 90 στην, ε, στην ομοθεσία της Ουγγαρίας. Απλώς η διαφορά είναι ότι τώρα γίνονται ιδεολογικές διαδηλώσεις από την κυβέρνηση και αυτό είναι προβληματικό. Για την περίπτωση του Αχμετ Έικ. Εμείς δεν σχολιάσαμε για την πρωτόβαθμη απόφαση Τη ε, πρωτοβαθμίας δίκη, αλλά για τον τρόπο που διεξάχθηκε η δίκη στο δικαστήριο, ε, όπου ε, οι κυβερνητικοί παράγοντες επηρέασαν την κατάσταση, υπήρξε απόλυτη δυνατότητα να προβλέψουμε κανείς ότι θα ακούγαμε ε, τιμιγορία ε, κατηγορίας. Από την άλλη, ναι, ε, στα σύνορα, παρότι Τραυματίστηκαν 300 ε, άτομα ε, από την άλλη μεριά ε, των συνόρων και παρότι κάποιοι αστυνομικοί επίση τραυματίστηκαν, δεν έγινε καμία σοβαρή έρευνα. Δεν αμφισβητούμε καθόλου ότι έριξε πέτρε ο κύριο αυτό και ότι χρησιμοποίησε μεγάφωνο, αλλά δεν μπορεί κανεί να χαρακτηρίσει τέτοιε πράξει ω τρομοκρατικέ πράξει. Υπάρχουν άλλα, άλλοι χαρακτηρισμοί πολύ πιο σωστοί και θα θέλαμε να απορριφθούν αυτέ οι κατηγορίε. Ο κύριος Σάντο. Ε, παρακαλώ, θα ήθελα να μιλήσω στα αγγλικά επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, γι' αυτό βάλτε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ. Εφτά άτομα είναι αυτά που ασχολούνται με, στην, στην Επιτροπή με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ, μαζί με άλλους δύο συναδέλφους, κάνω τις αναλύσεις. Ε, κυρία Σίπελ, δεν καταλαβαίνω γιατί σας ενδιαφέρει ποιος είναι ο αριθμός ε, του προσωπικού ή του κέντρου μας. Τα περισσότερα σχόλια που ακούστηκαν εδώ εμπνέονται από διάφορες ιδεολειψίες, ευχολόγια κτλ. Νομίζω ότι η σύμβαση της Γενέβης δεν εξασφαλίζει κοινωνικές παροχές. Μιλάμε για προσωρινή προστασία. Μόνο προσωρινή προστασία δίνει. Στην πρώτη ε, χώρα που μπαίνει κανένα. Παραδείγματο χάρη, ένα Σύριο πάει στη Λιβύη, α πούμε. Εκεί του πρέπει να το εξασφαλίσει αυτή η προστασία και όχι στην ε, Ουγγαρία. Ξέρω ότι δεν θα σα ευχαριστήσω. Για την υπόθεση Αχμέτα, θα σα δυσαρεστήσω. Συμφωνώ με τον πρόεδρο Ντόναλτ Τραμπ ότι ένα έθνος όταν δεν έχει σύνορα δεν είναι έθνος πια. Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από την προστασία των συνόρων. Δεν μπορούμε να ζητάμε λογαριασμό από ένα κράτος που θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του και γιατί ε, εκφράστηκε... Ε, και γιατί ελήφθη μία απόφαση πρώτο σε δικαστήριο. Από τη δεκαετία του 80 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η διεθνής κοινότητα ήταν συνηθισμένη σε φιλελεύθερα μέσα ενημέρωση στην Ουγγαρία. Σήμερα η κατάσταση όμως δεν είναι η ίδια, δεν είναι αυτή που είχαμε γνωρίσει στην αρχή της δεκαετίας του 2000. Ε, είναι πιο ισορροπημένη η κατάσταση. Έχει αλλάξει η αγορά και επομένως ε, αλλάζουν και οι απόψεις που εκφράζονται. Υπάρχουν πάρα πολλές επίσης οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών Ορισμένες ασχολούνται με θέματα πολιτική άλλε με κάτι άλλο. Τον υπόλοιπο χρόνο ο κύριο Τουτσάνη. I would like to Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να απαντήσω στα Ουγγρικά. Κυρίες ε, και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τα ερωτήματα που θέσατε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της κοινωνίας, ε, τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στην ε, Ουγγαρία έχουμε δημοκρατία. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε είδους διάλογο ή συζήτηση. Είναι φυσιολογικό αυτό. Υπάρχει κάτι όμως που με θλίβει. Αυτό που με θλίβει είναι ότι όταν μιλάμε για μετανάστευση δεν κάνουμε καμία διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Όλοι μιλάνε για πρόσφυγες κατά την άποψή μου. Η κατάσταση είναι πολύ πιο πολύπλοκη. Πρόκειται για μετανάστευση. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες μετανάστευσης που γνωρίζουμε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, οικονομικών μεταναστών. Οι οικονομικοί μετανάστες θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη από το Μαρόκο ή από άλλες χώρες για να ζήσουν καλύτερα από ό,τι στην πατρίδα τους. Δηλαδή από τη μία πλευρά υπάρχουν οικονομικοί μετανάστες και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι πρόσφυγες. Κανένα σήμερα δεν έκανε αυτή τη διάκριση. Παρόλα αυτά είναι μια πολύ σημαντική διάκριση και θα πρέπει να γίνεται. Με τον πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία, η Ουγγαρία επέδειξε ιδιαίτερη αλληλεγγύη. Η Ουγγαρία φιλοξένησε πάρα πολλούς ανθρώπους από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Έχουμε την τάση να ξεχνάμε, να ξεχνάμε την βοήθεια που έδωσε η Ουγγαρία σε αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης τίνουμε να ξεχνάμε το τι συνέβη το 1956 όταν πολλοί Ούγγροι πήγαν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να έχουμε απόλυτη συνείδηση του γεγονότος ότι οι άνθρωποι αυτοί συνεργάστηκαν με τις ε, αρχές. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Πάρα πολλοί, οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στην ίδια χώρα και γι' αυτό το λόγο η συνεργασία εδώ μετράει πάρα πολύ. Αυτό συμβαίνει το 2015. Όσοι φτάνουν στην Ουγγαρία δεν έχουν τελικό προορισμό την Ουγγαρία. Ο τελικός τους προορισμός είναι η Δυτική Ευρώπη, η Σουηδία κτλ. Παρόλο που έχουμε πάρα πολλούς εμπειρογνώμονες, πάρα πολλούς ειδικού. αν λάβουμε υπόψη μας τα στατιστικά δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν 9.000 εμπάλωτα άτομα που πέρασαν στην ε, Ουγγαρία πέρσι. Από αυτούς αυτές 9.000, οι 8.000 δεν περίμεναν το τέλος της διαδικασίας, αλλά αναχώρησαν για να πάνε στην Αυστρία ή τη Γερμανία τι θα πούν οι, οι ομολογοί μας ε, στην, στην ε, ε, Αυστρία. Θα μας πούν ότι θα πρέπει να προσφυλάξουμε καλύτερα τα σύνορά μας. Εγώ έζησα τη νεότητά μου σε καθεστώς κομμουνιστικό και εγώ ξέρω ότι παίρνει ε, δεν μπορεί κανείς ε, να πάρει το αυτοκίνητο και να οδηγήσει μέχρι τις Βρυξέλλες χωρίς να ελέγχεται. Δεν μπορούσε να το κάνει στο παρελθόν, μπορεί να το κάνει τώρα. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αφήσουμε να διακυβευτεί πάλι. Ε, αν πάτε στα σύνορα μεταξύ Αυστρίας και Ουγγαρίας θα δείτε τις πελώριες ουρές που υπάρχουν εμείς οι Ούγγροι ε, πρέπει να προφυλάξουμε τα εξωτερικά μας σύνορα για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε την ελευθερία διακίνησης. Όταν μιλάμε για μετανάστευση, ας κάνουμε μία προσπάθεια να δούμε τι ακριβώς ε, γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Πάρα πολύ λίγοι μεταφέρθηκαν αλλού από τους 160.000 και συγκεκριμένα 10.000. Μπορείτε βεβαίως εσείς ε, να κρίνετε, ε, μπορούμε, ε, ζητείτε να, η καταβολή 200.000 ευρώ προς τίμου εάν δεν δεχτεί, αν δεν δεχτούμε κάποιον. Αυτό είναι μια προσβολή για την κεντρική Ευρώπη. Θα πρέπει να πούμε την αλήθεια, θα πρέπει να σεβόμαστε τις διαδικασίες πάντοτε σεβαστή με τους νόμους στην Ευρώπη πάντοτε γινόταν έλεγχος, νομικός έλεγχος, δικαστικός έλεγχος, πάρα πολλές φορές τα ίδια τα δικαστήρια τροποποίησαν αποφάσεις που αφορούσαν θέματα ασύλου. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε μέτρα προκειμένου να προφυλάξουμε το χώρο Σέγγεν. Εμείς σεβαστήκαμε τα κριτήρια θα δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τα κοντέινες. θα ασχοληθούμε με τα παιδιά, αλλά όλα αυτά θα τα καταφέρουμε μόνον εάν γίνει σεβαστή η δημόσια τάξη και η δημόσια ασφάλεια. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Η τρομοκρατία τια βρίσκεται παντού, είναι πανταχού παρούσα. Δεν ξέρουμε ποτέ πού θα χτυπήσει η τρομοκρατία. Από ότι ε, γνωρίζω 14 Ιουλίου στην πρεσβεία, μάλλον στην πρεσβεία της Γαλλίας, μίλησα και είπα ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα επόμενα θύματα της τρομοκρατίας. Αυτό το είπα στις 14 Ιουλίου, στην Πρεσβεία το ίδιο βράδυ έγινε η επίθεση στη Νίκια. Η Κροατία, η Σλοβενία ε, έχουν κλείσει τα σύνορά τους και αυτά, αυτό δεν προκάλεσε τέτοιο σάλο όπως το κλείσιμο των δικών μας σύνορων. Όταν η Ισπανία έκλεισε τα σύνορά της για να ε, προφυλακτεί από τους Αφρικανούς ε, πρόσφυγες ε, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δεν εξανέστησαν τόσο πολύ. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή κρίση. Θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σε αυτή την κρίση και, επαναλαμβάνω, να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ μεταναστών και προσφύγων. Οι νέοι κανονισμοί που θα εισαχθούν θα είναι αυστηροί θα ορίσουμε υπεύθυνου στις κοινότητες και θα διεξάγεται ένας ε, έλεγχος, ένας αυστηρός έλεγχος. Και βεβαίως μπορεί ο καθένας να προσφύγει στο δικηγόρο του, εάν έχει κάποια διαφωνία. Θα ήθελα βεβαίως, και καταρχάς, να ασχοληθώ με τους ΜΚΟ. Πέρσι, όταν υπέβαλα ένα νομοσχέδιο που έδινε τη δυνατότητα στους ΜΚΟ να αναπτύξουν αμέσως δράση, κανένας ε, δεν με συνεχάρει. Είπαμε ότι η εγγραφή των ΜΚΟ θα έπρεπε να γίνεται αυτόματα, γιατί αυτό επέτρεπε την εύρυθμη λειτουργία τους. Κανένας ε, δεν με συνεχάρει. Δεν ζητάω συγχαρητήρια. Εγώ απλά και μόνο ζητάω αντικειμενικότητα γιατί αυτή η ε, εγγραφή ε, διευκόλυνε τα πράγματα. Υπάρχουν 60.000 ΜΚΟ στην Ουγγαρία. Βεβαίως είναι φυσιολογικό να υπάρχουν οργανώσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες. Είναι λογικό σε μια δημοκρατία. η κυβέρνηση έχει νομιμοποιηθεί μετά από τις εκλογές. Ε, ε, οι ΜΚΟ μπορούν να εκφράζουν ε, την άποψή τους. Όταν όμως δεν επιτρέπεται σε κάποιον να πει τη γνώμη του, θα πρέπει αμέσως να ακούγονται φωνές ότι πρόκειται για μια δικτατορία. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ΜΚΟ στο μέλλον, εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας. Εξέτασα την έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας θα νομοθετήσουμε για θέματα που είναι απόλυτα σαφή, θα πρέπει να υπάρχει εγγραφή τους στα ε, μητρώα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι, από πού έρχονται. Όλα αυτά είναι σύμφωνα με την έκθεση της Βενετίας και σύμφωνα με το πνεύμα της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει τίποτα που θα πρέπει να τους φοβίζει, να μην ανησυχούν λοιπόν. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για το θέμα των φυλακών. Ότι έχουμε πολλούς τρόφιμους στις φυλακές. Συζητήσαμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης το θέμα αυτό. Έχουμε επανεξετάσει 6.000 περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα από τα δικαστήρια, ε, έχουμε αλλάξει τις διαδικασίες και θα είναι πιο αποτελεσματικά, αποτελεσματικές. Ε, το Συνταγματικό Δικαστήριο επίσης μπορεί να ακυρώσει αποφάσεις των δικαστηρίων για το θέμα των τροφίμων. Ε, το Συνταγματικό Δικαστήριο λειτουργεί πάρα πολύ καλά και μάλιστα ακύρωσε και ένα νομοσχέδιο το οποίο το είχα κατεβάσει εγώ ίδιος. Αφορούσε την ε, μία νομική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση Αχμέντ, είπαμε πολλά, ακούστηκαν πολλά. Σε καμία περίπτωση όμως εγώ δεν θα ήθελα να κριτικάρω μία απόφαση ενός δικαστηρίου. Ποτέ δεν τόλμησα να πω ότι μία απόφαση δικαστική είναι καλή ή κακή. Ειδικά όταν δεν είναι τελεσίδικη. Ποτέ δεν πρόκειται να πω κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να εκφράσω καμία γνώμη για το θέμα αυτό. Μην περιμένετε κάτι τέτοιο. Ούτω ή άλλω υπεύθυνο είναι ο εισαγγελέα για την επαγγελία του κατηγορητηρίου και υπάρχουν και τα δικαστήρια στη χώρα. Και ο Υπουργό ε, Δικαιοσύνη δεν δικαιούται να πάρει θέση σε ό,τι αφορά μία απόφαση δικαστική. Θα ήθελα επίσης να πω δύο λόγια. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κύριος Νίντερ Μίλλερ για το θέμα των προσφύγων. Δεν ξέρω αν μιλάμε για την ίδια χώρα, έτσι. Αν υπάρχουν 200 ή 180 άτομα τα οποία θέλουν να περάσουν παράνομα από τα σύνορα, δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ε, μεταναστών ή προσφύγων στη Γαλλία Φερρυπίν. Υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα μου γιατί είχαμε πρόβλημα. Εγώ ήρθα σε επαφή με τον ε, Έλληνα πρόεδρο που είπε ότι κάθε μέρα 150 άτομα περνάνε την Τουρκία στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα από τη συμφωνία. Παρά τη συμφωνία με την Τουρκία περνάνε αυτά τα άτομα κάθε μέρα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα ενώ η Σερβία δεν είναι. Ε, τη στιγμή που είναι υποψήφια χώρα για την ένταξη, ε, τα κριτήρια της Κοπενχάγης εδώ πέρα υπάρχουν και θα πρέπει να τα σεβαστούν όλοι. Επίσης δεν φοβάμαι τις ΜΚΟ, ε, θέλω να υπάρχουν ΜΚΟ, συζητάω και στη Βουδαπέστη και αλλού με τις ΜΚΟ, φυσιολογικό είναι αυτό. Επίσης για τους νέους 14 με 18 χρονών νομίζω ότι οι αρχές θα μπορέσουν να διαχειριστούν το θέμα των νέων αυτών. Το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σχολιάσω αφορά το κομμουνιστικό καθεστώς. Φυσικά θα πρέπει να μιλήσουμε για τα κομμουνιστικά εγκλήματα, όπως πρέπει να μιλάμε και για το ολοκαύτωμα. Επίσης, θα πρέπει να μπορούμε να μιλάμε για εγκλήματα όπου και όποτε συμβαίνουν. Εμείς ε, ζήσαμε σε μια τέτοια χώρα με κομμουνιστικά εγκλήματα. Πρέπει να ενημερώσουμε τους νέους. Γιατί αν δεν τους ενημερώσουμε ε, δεν θα γνωρίζουν την ιστορία. Προσοχή όμως, ε, προσοχή, προσοχή με τους χαρακτηρισμούς περί δικτατορίας. Προφανώς θα πρέπει να μιλάμε για τα κομμουνιστικά εγκλήματα. Δώστε μου ακόμα δύο λεφτά σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ε, γυναικών και την σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης. Είμαστε σε φάση διαβούλευσης. Ε, θα δούμε τι θα προκύψει το Σεπτέμβριο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί ότι είναι θέμα προτεραιότητας η προστασία των θυμάτων, των γυναικών δηλαδή, και υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα εν το γεννάστε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις συνεισφορές σας. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Είμαι έτοιμος να συζητήσω. Μόνο έτσι μπορούμε να συζητάμε. Όσοι κάνουνε... Όσοι μιλάνε για το άρθρο 7 θα πρέπει αυτό να μην το δεχτούμε. Ε, το άρθρο 2 είναι σημαντικό για μένα ε, και για το δικαίωμα των παιδιών. Αυτή πρέπει να είναι η βάση για την ε, οικοδόμηση της Ευρώπης. Σίγουρα πρέπει να πούμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πλούσιες χώρες, ε, φτωχές χώρες, μεγάλες χώρες, μικρές χώρες. Χώρες που ήταν πριν το 2004, χώρες που μπήκαν μετά. Δεν είναι καλό αυτό. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Ε, για την ε, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη υπάρχουν διάφοροι νόμοι ε, που προωθούν τις διακρίσεις, ε, που προσπαθούν να βάλουν στο περιθώριο τις επιχειρήσεις. Ε, που δεν σέβονται το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ε, εγώ πάντως νομίζω ότι για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να υπάρξει διάλογος. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ο κύριος Μωράες. Πρόεδρε, ε, συνάδελφοι, θα πρέπει να κλείσουμε εδώ ε, αυτή την ακρόαση. Ο κύριος Βίστεσεν ε, αμφισβήτησε τη σημασία το κατά πόσο να έχει νόημα να φτιάξουμε μια τέτοια, να οργανώσουμε μια τέτοια ακρόαση. Ε, το σκεφτήκαμε πάρα πολύ σοβαρά. Είναι προνόμιο του Κοινοβουλίου να εξετάσει την ε, κατάσταση των δικαιωμάτων στην, ε, σε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ όλου όσου μίλησαν σήμερα. Ε, πέρασαν όλα τα μηνύματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του ομιλητέ και του πανελίστε. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να απαντήσουν ε, πολύ βαθίε ερωτήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολύ ενδελεχείς, πολύ λεπτομερεί. Καμία ακρόαση δεν είναι τέλεια, αλλά ευχαριστώ όλου όσου συμμετείχαν και που συνεισέφεραν τόσο ώστε να είναι στον δόν πιο ισορροπημένοι. Τώρα κλείνουμε αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ την ακρόαση. Ε, θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες στις 5. Παρακαλώ να είσαστε εδώ στις 5 για να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Good afternoon, colleagues. We can begin the vote whenever... Καλησπέρα συνάδελφοι, μπορούμε να αρχίσουμε όταν είστε έτοιμοι, παρακαλώ καθίστε. Δεν έχουμε εκτός από τις ψηφοφορίες κανένα άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη, γι' αυτό και μπορούμε πιστεύω να τα τελειώσουμε όλα στην ώρα τους. Είμαστε όλοι έτοιμοι, οι συντονιστές, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, αν κάποιο δεν έχει την ηλεκτρονική του κάρτα, ας μας κάνει ένα σήμα. Τότε θα πάρουμε την ψήφο σας διανάτασης της χειρός. Οπότε όλοι έχουμε ηλεκτρονικές κάρτες. Ναι. Αν είμαστε όλοι έτοιμοι μπορούμε να αρχίσουμε με την πρώτη ψηφοφορία, εντάξει. Έχουμε τον κύριο, την κυρία Στίβενς τώρα, αντί της οποίας είναι ο κύριος Σκρίπεκ. Κανείς από τους δύο είναι εδώ. Είναι κάποιος από το ECR εδώ σήμερα. Αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ναι, μπορούμε. Κανείς δεν θέλει τον λόγο, τέλεια. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 12. Συγγνώμη, τι ψηφίζουμε. Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν επί βατηγά πλοία λοιπά. Έναρξη ψηφοφορία. Τροπολογία 12. Έκλεισε. Εγκρίθηκε. Ο κύριος Κρύπας κάθεται. Ας του παραδώσουμε την άξιο. Πρέπει να καθίσει μερικά λεπτά δευτερόλεπτα, συνάδελφοι. Θα περιμένουμε τον κύριο Σκρίπεκ να καθίσει. Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτό, είστε έτοιμοι. Τροπολογία 13. Άνοιξε. Πέρα στις ψηφοφορίες. 14, τροπολογία 14, έναρξη, πέρας, εγκρίνεται, 15, έναρξη, πέρας, εγκρίθηκε, 17, έναρξη, πέρας, απορρίφθηκε. 16, τροπολογία 16, έναρξη. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 18, έναρξη. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 19, έναρξη. Πέραση ψηφοφορίας απορρίφθηκε τροπολογία 21, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας, απορρίφθηκε. Τροπολογία 21 έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, εγκρίθηκε. Τροπολογία 22, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, Εγκρίθηκε τροπολογία 23, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε αιτιολογικές σκέψεις, ένα, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 2, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας απορριφθήκε. Τροπολογία 3, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, απορριφθήκε. Τροπολογία 4, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, απορριφθήκε. Τροπολογία 5, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, εγκρίθηκε. Παρόλο αυτό που προέκυψε στην οθόνη, η επόμενη τροπολογία, η έκτη, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, απορρίφθηκε. Έβδομη τροπολογία, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, απορρίφθηκε. Τροπολογία 8. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 9. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 10. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 10. Συγγνώμη, τροπολογία 11. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας απορριφθήκε. Συνάδελφοι λοιπόν, σύμφωνα με τον κανόνα 544, τώρα θα προχωρήσω στην παρουσίαση των τροπολογιών εκ μέρους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε τώρα στην εφαρμογή της δεγόμενης αποφασής πριν από τα κράτη-μέλη. Ζητήθηκε η γνώμη του Κοινοβουλίου για τους φακέλους αυτούς εντός τριών μηνών. Τέλος των διαβουλεύσεων ήταν 23 Φεβρουαρίου. Ζητήσαμε μια παράπαση της προθεσμίας υπάρχει στα αγγλικά μόνο. Η έκθεση παρουσιάστηκε στην συνεδρίασή μας της 9 Φεβρουαρίου. Δεν προτάθηκαν τροπολογίες, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, η οποία θα γίνει στην Ολομέλεια τον Μάρτιο, οπότε αν είστε έτοιμοι για την ψηφοφορία μπορούμε να προχωρήσουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε με 42 ψήφους υπέρ, 2 κατά. Οπότε πάμε στο επόμενο. Πάλι στη λεγόμενη απόφαση πριν. Υπενθυμίζω και πάλι τα ίδια που ισχύουν και για την προηγούμενη τροπολογία. Διαβουλεύσεις έως 23 Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε στις 9 Φεβρουαρίου, γι' αυτό και προχωρούμε και πάλι στην ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, εγκρίθηκε. Περνάμε στο σημείο 7. ψηφοφορία για τη θέσπιση ενός συστήματος εισόδου-εξόδου για την καταχώρηση δεδομένων εισόδου και εξόδου, καθώς και άρνηση εισόδου ειδικών τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορισμός των όρων πρόσβασης στο σύστημα εισόδου-εξόδου για σκοπούς επιβολής του νόμου. Ο εισηγητής έχει τον λόγο. Κύριε Ντιάζ Ταμέρα, θέλετε τον λόγο. Εν συντομία, κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλώς να ευχαριστήσω όλες ε, τις πολιτικές δομάρτες που δούλεψαν τόσο σκληρά. Ευχαριστώ. Είστε έτοιμοι για την ψηφοφορία, Ηνωμένο Βασίλειο. Ωραία, χαίρομαι που το ΕΛΚ είναι εντάξει Ωραία. Πάντοτε ευχάριστο αυτό. Τροπολογία 149, 151, 152, 3. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται Τροπολογία 154. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός. 1. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός και άρθρο 1. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός και άρθρο 2. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 333, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Συμπεριβασμός και άρθρο 3, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας, εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 353. Τροπολογία. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 3-5-4. Έναξη. τρία πέντε τέσσερα εναξη περας απορριπτεται Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο 6. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η κυρία Σπινέλη απέχει. Α, δεν λειτουργεί το μηχάνημά της μπροστά. Θέλετε να αλλάξετε θέση, κυρία Σπινέλη. Μισό λεπτό. Έτοιμοι. Συμβασμός και άρθρο 9. Ωραία. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε το 39. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός. Α, δύο 3, 9, 9, 2. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Σύπιος και άρθρο 9. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο 10. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέσσερα δεκατέσσερα. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τέσσερα ένα πέντε. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 41, έναξι, πέρας, εγκρίνεται. 417, έναξι. Τέσσερα είναι επτά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Έναρξη. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Έναρξη. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός και άρθρο 12. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Σύμβασμός για το άρθρο 13. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Σύμβασμός για άρθρο 14. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός και άρθρο 15, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός και άρθρο 16, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός. Τροπολογία 4 Τροπολογία 4-6-5. έναρξη της ψηφοφορίας. 4-6-5 ψηφίζουμε. Πέρας φιγουρίες. Εγκρίνεται συμβασμός και άρθρο 17. Πέρας. Εγκρίνεται συμβασμός και άρθρο 15. Έναξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο 19. έναξι, Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο 20. Έναξη. Πέρας. Εγκρίνεται συμβασμός και άρθρο 21. Έναξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμό στο κεφάλαιο 3, άρθρα 22-25. Έναξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 5-19. Έναξη. Πέρας. Απορρίπτεται κεφάλαιο 4. Έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες. 5-30 τροπολογίες. Έναξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός και άρθρο. Τροπολογία 5.33. Έναρξη ψηφοφορίας. 5.33. Τροπολογία. Πέρας. Απορρίπτεται. 5.34. Έναρξη. 5.34. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός και άρθρο 31. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός και άρθρο 32. Έναρξη. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο 33. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο 34. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο... Μισό λεπτό. Προπολογισμός 17. Α, 16, 16, έναρξη. Έναρξη ψηφοφορίας. υπολογισμό 16. Έναρξη ψηφοφορίας. Προπολογισμός 16. Πέρας. Εγκρίν. Απορρίπτεται. Συμβιβασμό και άρθρο 35. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμό για το άρθρο 36. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται συμβασμός και άρθρο 37. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός και άρθρο 38. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τοπολογία 636. 636. Ψηφίζουμε. Πέρας απορρίπτεται. 6.38 έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός και άρθρο 39 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Σειρά από τεχνικές ε, τροπολογίες ομάδα τροπολογιών. Πέρας φιουφορίας εγκρίνεται. Δε... 105-107 σύνολο τροπολογιών, ομάδα τροπολογιών. Περνάμε στο συμβιβασμό και το άρθρο 40. έναξι, πέρας, εγκρίνεται. Τροπολογία 84, έναξι, πέρας, εγκρίνεται. 85, έναρξη, πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο 44. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 6-4-1. Έναρξη. Πέρας. Τροπολογία 95. Έναρξη. Θα πρέπει να ψηφίσουμε προσεκτικά έναρξη, πέρας, εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο 46. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. έξι τέσσερα Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. πέντε Έναρξη. Συνάδελφοι, η τροπολογία συν 665 υπάρχει ένας συνάδελφος από το ΕΛΚ που περισσεύει. Μήπως θα μπορούσε να αποσυρθεί ένας συνάδελφος. Θα μπορούσε, θα μπορούσε κανείς να αποσυρθεί. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Επεσύρθη κάποιος. Ωραία, 665 πάλι. Ευχαριστώ Ρομπέρτο. Πέρας. Εγκρίνεται. 104 ψηφίζουμε τροπολογία. Πέρας. Εγκρίνεται. 106. 106, Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 666. Α, αυτή είναι του διαβόλου. Η Ρεβέκα μου το είπε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο 49. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο 50. Έναρξη. Ελπίζω να περάσει αυτή. Α, κανένα δεν το στο αστείο. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ωραία, ωραία. Τροπολογία 671. Έναρξη. Πέρας απορρίπτεται. Συμβασμός για άρθρο 51. Έναρξη. Εγκρίνεται. Συμβασμός και άρθρο 52. Έναρξη. Πέρας. Δεν πειράζει, εντάξει, έναρξη. 53. Εγκρίνεται. Σύμφασμός και άρθρο 54, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός και άρθρο 55, έναρξη. Πέρας. Carried. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός επί του άρθρου 56. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική επί του άρθρου 57. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας εγκρίνεται. Συμβιβαστική επί άρθρου 58, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική επί άρθρου 59, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική επί άρθρου 64, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 720, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 142, έναρξη ψηφοφορίας, Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 721. Έναρξη ψηφοφορίας. Τάνια, θέλεις, θέλεις να πεις κάτι. Αν και στις τροπολογίες δεν λέμε συνήθως κάτι, συγγνώμη, αστείο ήταν, αστείο ήταν. Είναι Δευτέρα και έχω αυτή τη διάθεση. Λυπάμαι, ήταν ένα αστείακι. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Είναι, μπορεί να σχετίζεται με την Ουγγαρία, δεν ξέρω. Δεν θα πω ό,τι θέλω να πω, αλλά είμαστε στην 721, όπου έχω μια προφορική τροπολογία, οπότε προχώρησε. Ευχαριστώ. Θα τη διαβάσω. Η παράγραφο 2 θα ισχύει επί δύο χρόνια από την αρχή της λειτουργίας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 και όχι, μετά και όχι πριν από μια έκθεση αξιολόγησης και αποστολή της στο Κοινοβούλιο έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορατότητα και η αναγκαιότητά της. Ευχαριστώ πολύ Τάνια. Ας ψηφίσουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Περνούμε στις παραπομπές, έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, εγκρίνεται. Τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Οπότε περνάμε επιτέλους στην τελευταία ψηφοφορία. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Είμαστε όλοι έτοιμοι τελική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται με 46 υπέρ 38 κατά μία αποχή. Τα συγχαρητήριά μου κύριε Διάς Γαμέρα. Κυρία Βέζια, θέλετε τον λόγο. Ναι, παρά την ε, υιοθέτηση δύο από τις τροπολογίες μου, η Γκουε θέλει να καταθέσει ψήφισμα μειοψηφία για να εξηγήσει την ψήφο με βάση το άρθρο 52 παράγραφος 4, ε, κύριε Πρόεδρε. Αποδεκτό. Κύριε, κύριε Ντίας Δεμέρα, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όχι. Ζητώ συγγνώμη. Πρόεδρε. Κύριε Ντίας Δεμέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η κυρία Βεργιά έχει απόλυτο δίκιο να χρησιμοποιήσει το 52α. Ε, είναι το δικαίωμα της ε, μειοψηφίας. βάση τα δικαιώματα που έχει η μειοψηφία μπορεί να κάνει επίκληση αυτού του άρθρου. Το σέβομαι. Το περίμενα κύριε στα Στεμέρα προφανώς. Ε, συνάδελφοι, τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε με βάση το άρθρο 69C την τελική ψηφοφορία για την απόφαση να γίνουν διαπραγματεύσεις ε, την σύνθεση ε, Βουλής, παράγραφος 69β και 69γ. Ψηφίσουμε τώρα. Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. 4 ψήφοι υπέρ, 40 ε, ψήφοι συγγνώμη, υπέρ, 4 ψήφοι κατά, μία α, αποχή. Συγχαρητήρια και πάμε τώρα πάλι στο κείμενο του κ. Ντία Δεμέρα, πριν περάσουμε στην ψηφοφορία. Θέλετε, κ. Ντία Δεμέρα, να πάρει το λόγο. Τότε πάμε στην ψηφοφορία απευθεία. Τροπολογίε 20, 21 και 22 μαζί. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική 1. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία έτσι ώστε να χαρούμε όλοι μας έναρξη ψηφοφορίας ονομαστική. Εδώ, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, για να σας κάνω ευτυχισμένους. Τελική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίες, εγκρίνεται με 38 και 7 ψήφους, κατά και αποχές αντίστοιχα. Κυρία Μπερζιά, Αλλάξατε γνώμη αυτή τη φορά. Όχι, δεν άλλαξα γνώμη. Αυτή η έκθεση όμως είναι απόρρια της προηγούμενης. Επομένως, ε, αρκεί μία φορά το ψήφισμα αυτό μειοψηφία. Αρκεί, δεν χρειάζεται και δεύτερο. Πολύ ωραία. Ισχύει και για αυτή, λοιπόν. Λοιπόν, σύμφωνα με το 69C, έχει αρχίσει, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με έναν και τέσσερις ψήφους κατά και μία αποχή. Η έκθεση θα κατατεθεί στην Ολομέλεια στις 2 Μαρτίου. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Είναι το τέλος αυτό. Ναι, είναι το τέλος της ψηφοφορίας και το τέλος της συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για την προσοχή σας σήμερα.